Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, λειτουργεί το μικρόφωνο μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε όμως τον πρόεδρό μας, ο οποίος βρίσκεται σε μια άλλη συνεδρία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προεδρεύσω για το πρώτο μισό του απογεύματός μας. Και ξεκινώντας την απογευματινή συνεδρίαση, έχω την τιμή και τη χαρά να καλωσορίσω τον πρεσβευτή της Νορβηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Άντλε Λάικβολ. Πριν από δύο χρόνια κύριε Πρεσβευτά είχαμε την τελευταία ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τότε είχαμε κάποια προβλήματα στην ημέρηση διαταξή μας τα οποία μας απασχόλησαν ιδιαίτερα. Παραδείγματος χάρη οι δασμοί για τα δρεπτά άνθη και επίσης οι δασμοί για κάποια είδη κρέατος και τυρού. Όλα αυτά οδήγησαν σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2013 σε σχέση με την αύξηση των δασμών για αγροτικά προϊόντα. Τα χρόνια περνούν και δεν ξαναγυρίζουν. Με τον τρόπο όμως αυτό υπήρξαν και πολλές αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε εμπορικό επίπεδο. Και η Νορβηγία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς και τους εξαγωγούς τους έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο. Λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι προσπάθειες λοιπόν φιλελευθεροποίησης μεταξύ των οποίων και αυτά τα προϊόντα τα αγροτικά που υπόκειται στο άρθρο 19 της Συμφωνίας Ελεύθερου Οικονομικού Χώρου ε, πρέπει να προχωρήσουμε στη φιλελευθερωποίησή του. Είναι πιο επίγον από ό,τι ποτέ. Κύριε Πεσβευτά, λοιπόν, θα σα δώσω το λόγο και φυσικά και η Κομισιόν μπορεί να λάβει το λόγο στη συνέχεια και θα ακολουθήσουν τα ερωτήματα των μελών. Εξοχότατε, λοιπόν, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σα και ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Όπως είπατε, ε, έχουν περάσει δύο χρόνια από την προηγούμενη πρόσκληση που μου απευθύνθηκε. Βλέπω ένα νέο κοινοβούλιο με, πολλά, με πολλά παλιά πρόσωπα αλλά και πολλά καινούργια πρόσωπα. Πάλι σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση να συζητήσουμε τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας συμπεριλαμβανομένων και των προοπτικών για περαιτέρω φιλελευθεροποίηση στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Θα είμαι σύντομο. αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω μια γενική εικόνα χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη περίπτωση. Τέσσερα λοιπόν σημεία θέλω να υπογραμμίσω. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν για τη γενική εικόνα, δεύτερον για τα ενεργειακά θέματα, τρίτον για τα, την αλληλεία και το τέταρτο μονάχα για τη γεωργία. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσω να εξασφαλίσω τη δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούμε να έχουμε μια καρποφόρα και επικοδομητική συζήτηση για το, τη γενική εικόνα. Η Νορβηγία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έβδομη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη. 75% τα τρία τέταρτα των εξαγωγών μας, του συνολικού μας εξωτερικού εμπορίου, πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τεράστιο και δείχνει το βαθμό ολοκλήρωσης και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και φυσικά δείχνει και τα αμοιβαία ωφέλη που προκύπτουν. Πέραν όμως του εμπορίου δείχνει την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Αν εξαιρέσουμε τους πρωτογενείς παράγοντες, η Νορβηγία έχει το διεθνιστικό πλαίσιο όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την συμφωνία του ΕΟΧ, η Νορβηγία είναι τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Έχουμε ακριβώς το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα αγαθά της υπηρεσίας, το κεφάλαιο και τα άτομα και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Horizon 2020 Ιεράσμος ΣΥΝ και άλλα προγράμματα. Έχουμε ξεπεράσει τώρα το επίπεδο του 10.000. 10.000 νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενσωματωθεί στο νορβηγικό δίκαιο. Αυτό δείχνει το πόσα πράγματα καλύπτει η ενιαία αγορά και πόσο σημαντική είναι η συμφωνία του ΕΟΧ 20 χρόνια λοιπόν έχουν περάσει και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια αυτό το πλαίσιο αποδείχθηκε δυναμικό και ανθεκτικό. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι η οικονομική ολοκλήρωση και όχι μονάχα οι εμπορικές σχέσεις, το ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και το αμοιβαίο κέρδος. Δεύτερο σημείο, η ενέργεια. Είναι μεγάλα τα στοιχεία του εμπορίου μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 20% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% του πετρελαίου προέρχονται από την Νορβηγία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα τη οικονομική ολοκλήρωση. Έχουμε το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο και έχουμε και μια εταιρική σχέση. Η Νορβηγία είναι ένα σταθερό πάροχο ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι μονάχα οι εξαγωγέ των ενεργειακών προϊόντων, τα αμοιβαία ωφέλη. 40% από την υφαλοκρηπίδα της Νορβηγίας ε, ελέγχονται από ευρωπαϊκές εταιρείες και η δραστηριότητά τους αφορά 100.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν εμείς συζητούμε τα ενεργειακά θέματα και την κλιματική αλλαγή, τα θέματα της ενεργικής αποδοτικότητας και την ασφάλεια εφοδιασμού και τα θέτουμε στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντα, αυτή η εταιρική σχέση είναι πιο σημαντική από ποτέ στο παρελθόν. Τρίτο σημείο, τα θαλασσινά και η αλία δεν καλύπτεται από τις γενικές ε, πρόνοιες του ΕΟΧ. Οι νορβηγικές εξαγωγές έχουν να αντιμετωπίσουν εμπορικά, εμπορικούς φραγμούς και δασμούς στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα θέλαμε να αρθούν αυτοί οι φραγμοί και οι δασμοί, τουλάχιστον να μειωθούν. Παρ' όλα αυτά, τα εμπορικά στοιχεία, οι ροές εμπορικές είναι πολύ σημαντικές. 60% από τις συνολικές εξαγωγές μας πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι είχαμε συνολικές εξαγωγές 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για ε, προϊόντα αλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και πάλι υπάρχει το στοιχείο αυτό του αμοιβαίου ωφέλους. Κανονικά σας στέλνουμε πρώτη ύλη την οποία εσείς μετά επεξεργάζεστε. 12.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με τη μεταποίηση αλλιευτικών προϊόντων από την Νορβηγία. Είπατε κύριε Πρόεδρε ότι υπάρχει το πρόβλημα της ρωσικής στάσης και του εμπάρκου. Εδώ τονίζω τη σημασία του να έχουμε αλληλεγγύη όταν υπάρχουν αναταραχές σε γεωπολιτικό επίπεδο. Τα αλληλευτικά προϊόντα ήταν το πιο σημαντικό εξαγωγικό μας προϊόν προς τη Ρωσία. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μια αγορά πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ εξανεμίστηκε. Και αυτό σας δείχνει πόσο Σημαντικό είναι το ότι πρέπει να είμαστε μαζί σε πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνουμε και ένα τίμημα σε ό,τι αφορά τη ρωσική αγορά εξαγωγών μας για τα αλληλευτικά προϊόντα. Είναι τεράστια λοιπόν η αγορά αλληλευτικών προϊόντων. Θέλουμε να, βοηθήσουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά και είδαμε πόσο συνδέονται τα γεωπολιτικά προβλήματα και το εμπόριο. Τέλος η Γεωργία. Mm. Η γεωργία δεν καλύπτεται από τις γενικές ρήτρε του ΕΟΧ, το άρθρο 19. Γενικά η Νορβηγία εισάγει τα 50% της συνολικής της κατανάλωσης για προφανείς λόγους στον αγροτικό τομέα. Το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ εκτενές, πάνω από 60% μεταξύ 60% και 70% των συνολικών μας εισαγωγών έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η γενική εικόνα λοιπόν. Και αυτό με φέρνει στα συγκεκριμένα μέτρα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πριν από δύο χρόνια με προσκαλέσατε και ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο με προσκαλέσατε σήμερα. Μπορώ να σας διαβεβαίωσω κύριε Πρόεδρε ότι δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία σε σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας έχει γίνει σαφές. Για μένα είναι κάτι το οποίο ε, γνωρίζω μετά από διμερείς επαφές σε διάφορα επίπεδα, μετά από <laughs> επίσημες συνεδριάσεις όπως αυτές του Συμβουλίου του ΕΟΧ και επίσης και σε προηγούμενες επαφές μου με την Επιτροπή σας. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω σήμερα είναι απλώ να σας ενημερώσω για τρία στοιχεία. Πρώτα, τα πολιτικά στοιχεία. Όπως θυμόσαστε, υπήρξαν διαφωνίες και στην Νορβηγία όταν τα μέτρα αυτά εισήχθησαν. τα κόμματα που βρίσκονται τώρα στην εξουσία στην Νορβηγία τότε είχαν διαφωνήσει και θέλαν να ακυρώσουν τα μέτρα αυτά όταν ερχόντουσαν στην κυβέρνηση. Πέρσι πήραν πραγματικά τα κόμματα αυτά στην εξουσία. Θέλαν να ακυρώσουν αυτά τα μέτρα αλλά τόνισαν εφόσον η κυβέρνηση μειοψηφία ότι χρειαζόταν την σύμφωνη γνώμη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου για να το κάνουν. Και δεν πήραν αυτή την υποστήριξη. Τρίτο στοιχείο είναι το ουσιαστικό εμπόριο. Τι έχει γίνει σε επίπεδο πραγματικού εμπορίου. Αν δούμε τα στοιχεία για το 2013-2014, βλέπουμε ότι τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στα μέτρα αυτά, η αλλαγή από ειδικού δασμούς σε δασμούς ad οδήγησαν σε ένα επίπεδο δασμών που είναι περίπου το ίδιο από αυτό που ισχύει προηγουμένως. Μια μικρή μείωση το 2013, μια μικρή αύξηση το 2014 για το εμπόριο. Δεν άλλαξε ουσιαστικά το επίπεδο του εμπόριου. Και ένα περαιτέρω στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα των διαπραγματεύσεων. Στη συμφωνία του ΕΟΧ, που είναι η πληρέστερη συμφωνία στην οποία έχει ε, δεσμευτεί η Νορβηγία το άρθρο 18 λέει ότι θα πρέπει τα συμβαλόμενα μέρη να συνεχίσουν τις προσπαθίε του ώστε να υπάρξει προοδευτική φιλελευθερωποίηση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων μέσα στο πλαίσιο τη αγροτική του πολιτική και επίση θα πρέπει να το κάνουν με έναν τρόπο που να είναι αμοιβαία επωφελής. Η Νορβηγία εδώ και πολλού μήνε τόνισε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τα αγροτικά προϊόντα επί τη βάση των ρητών του άρθρου 19. Εγώ έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στις διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να φιλελευθερωποιήσουμε ακόμα περισσότερο το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν κύριε Πρόεδρε, υπομορφή εισαγωγή. Έχουμε κάποιε μεγάλε προοπτικέ, έχουμε σημαντικού τομεί που εμπλέκονται στο εμπόριο. Το πιο σημαντικό όμω είναι η οικονομική ολοκλήρωση. Τα αποτελέσματα επίση των γεωπολιτικών διαταραχών στο εμπόριο και τέλος αυτά τα οποία μπορώ να σας πω για τα ειδικά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν τον Ιανουάριο του έτους αυτού. Και προσβλέπω σε μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρεσβευτά για αυτά που μας είπατε που ήταν πολύ καλά δομημένα αλλά και οι συνάδελφοί μου εδώ νομίζω θα σας διατυπώσουν ερωτήματα. Πριν δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στην Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση της Γεωργίας να μας διατυπώσει μία σύντομη παρουσίαση. Κυρία Βαλενζουέλα, ως επικεφαλής της μονάδας αυτή, μιας μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έχει πολύ στενές γεωργικές σχέσεις με την Νορβηγία. Είναι η έβδομη εξαγωγική μας αγορά για τρόφιμα και βασικά γεωργικά προϊόντα. Οι σχέσεις αυτές αυξάνονται συνεχώς. Από 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πριν από μερικά χρόνια σε σχεδόν το διπλάσιο. Οι εξαγωγές μας γεωργικών προϊόντων ανέρχονται σε 8,1% των συνολικών εξαγωγών μας στην Νορβηγία. Παρά όμως το σημαντικό ύψος αυτού του εμπορίου υπάρχουν και δύο φραγμοί, δύο εμπόδια που παρεμποδίζουν τις γενικά καλές εμπορικές μας σχέσεις. Η Νορβηγία δεν έχει ακόμα αλλάξει καταργήσει την ταξινόμηση που αφορά μερικά τυριά και μερικά κρέατα πρόβια. Η Κομισιόν ζήτησε να ληφθούν και τα δύο αυτά μέτρα για σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο λέγοντας ότι θεωρεί την αντίθεση σε αυτούς, στην άρση αυτών των φραγμών σαν προστατευτισμό. Σαν ίδιο πνεύμα καλέσαμε την Νορβηγία να καταργήσει αυτά τα μέτρα αλλά παρά τα θετικά, τη θετική ανταπόκριση που είχαμε από την Νορβηγία μέχρι σήμερα δεν καταργήθηκαν αυτά τα μέτρα και γι' αυτό παρά το ότι δεχόμαστε την πρωτοβουλία τους να αρχίσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το άρθρο 90. Ελπίζουμε ότι ο γύρος αυτός θα αποτελέσει ένα πλαίσιο για να λυθούν αυτά τα δύο εκρεμή προβλήματα για να υπάρξει πραγματική απελευθέρωση του γεωργικού τομέα στο εμπόριο για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τα μέλη της Επιτροπής μας Πρώτα οι πολιτικές ομάδες. ΕΛΚ πρώτα ο συντονιστής Δανιέλ Ντεκάσπαρη. Να. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη για το γεγονός ότι δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε παρόν. Εγώ θέλω επίσης να σε ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε πάρα πολλούς τομείς. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσεις, κυρίως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την αλληλέγγυα στάση σα και φυσικά τονίσατε πόσο καλέ είναι οι σχέσει μα, αλλά φυσικά και οι δύο πλευρές αντλούν ωφέλη από αυτέ. Αλλά ήσασταν και παρόντε μαζί μα πριν από δύο χρόνια εδώ και εκφράσατε την, την ε, αντίρρηση μας στο γεγονός ότι υπήρξαν μέτρα που εισήχθησαν από την Ορτηγία χωρίς όπως προβλέπουν οι συνθήκες να υπάρξει διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράγραφος 19 ε, λέει ότι πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση του εμπορίου και όχι περιορισμός. Τα μέτρα τα οποία είναι ανδεκτά από την Ορβηγία είναι φανερό ότι περιορίζουν το εμπόριο με αυξήσεις στους δασμούς και τους φραγμούς. Παραγωγή χάρη αυτό αφορούσε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία οι δασμοί δεκαπλασιάστηκαν. Έχω λοιπόν δυσκολίες να δεχθώ αυτά τα οποία λέτε. Λέτε ότι θέλετε να βελτιώσουμε από τη μια μεριά τις σχέσεις μεταξύ μας. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησής σας έχουν επιδεινώσει την κατάσταση των διμερών μας σχέσεων και εγώ θεωρώ ότι πρέπει τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν οδηγήσει σε προβλήματα θα πρέπει να ακυρωθούν Πρωτού προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις και δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολα τα πράγματα όταν, θα, όταν δίνουμε στην Κομισιόν μια διαπραγματευτική εντολή και μας λέει η Κομισιόν πρέπει να διαπραγματευτούμε για πράγματα τα οποία έχουν ήδη αποφασιστεί εδώ και πολύ καιρό. Όχι λοιπόν μονάχα το ότι πρέπει να αρθούν αυτά τα νέα μέτρα τα οποία έχετε κάνει, αλλά πρέπει να γίνουν και νέες παραχωρήσεις αν θέλετε να έχουμε αυτή την φιλική σχέση. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάνουμε διαπραγματεύσεις χωρίς να ακυρώσετε αυτά τα μέτρα τα οποία μας έχουν δυσαρεστήσει στο παρελθόν. Είναι σαν να παίζετε με τη φωτιά. Είναι πολλοί συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν πολλές ε, αμφιβολίες για αυτά τα μέτρα αν στο φως αυτών μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται για περαιτέρω ε, διευκολύνσεις όταν είναι φανερό ότι έχουν παραβιαστεί οι ρήτρες της συμφωνίας του ΕΟΧ. Είναι μια πλειοψηφία λοιπόν των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι δυσαρεστημένα με αυτά τα μέτρα και αυτό θέτει σε κίνδυνο την περαιτέρω συνεργασία μας. David Μάρτιν από Πολύ σύντομα. Εγώ έχω λίγο διαφορετική θέση από τον Ντάνιελ και σέβομαι το γεγονός ότι η Νορβηγία είναι ανεξάρτητο κράτος και άρα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για τον λαό της Φαίνεται ωστόσο να το κάνετε χωρίς να λάβετε σοβαρά υπόψη τα προβλήματα των, των γειτόνων σας. Δηλαδή και η Κομισιόν έχει αυτή την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς με, ποιο, με ποιον κόσμο διπραγματεύεστε. Δηλαδή δεν αμφισβητούμε ότι έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αυτές τις αποφάσεις αλλά το αν λαμβάνετε υπόψη τις γνώμες των γειτόνων σας πριν λάβετε την απόφαση. Δηλαδή εσείς λαμβάνετε την απόφαση και μετά τη συζητάτε και μετά και δεν ασχολείστε με τη γνώμη των ε, γύρω σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσύ άρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβε, εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω κάποιες βασικές πληροφορίες όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν υπάρχει σχεωριστή συμφωνία για το τι ακριβώς συμβάλλετε εσείς προς την Ένωση. Από ό,τι κατάλαβα, για την, ε, κατά τη γνώμη της Νορβηγίας. Δηλαδή πόσο πληρώνεται για την πρόσβαση στην ενιαία αγορά και δεύτερον πόσοι από τους εθνικούς σας νόμους, την εθνική σας νομοθεσία αποτελείται από νομοθεσίες περί της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Είναι ενδιαφέρον και σημαντικό για τη συζήτηση και χρήσιμο να το γνωρίζουμε γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους. Η κυρία Σέκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ε, και ευχαριστώ, Πρέσβη. Συγγνώμη που σας γυρνώ την πλάτη, αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ καθισμένη. Μετά από όσα ήδη υπόθηκαν, εγώ θα ήθελα να εστιάσω λίγο περισσότερο στον αντίκτυπο ε, του εμπάργου της Ρωσίας ε, στην Ένωση και την Νορβηγία. έχει γίνει το εμπάργκο και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ε, για την εξόριξη πετρελαίου στην Αρκτική και θέλω θέλω να γνωρίζω ποιες είναι οι απόψεις του πρέσβη για τις επιπτώσεις του εμπάργου στον τομέα της ενέργειας και της ε, ε, ναυσιπλοείας. Υπήρξε, από ό,τι κατάλαβα, μια ερώτηση για το αν μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες σας μια σχετική, υπηρεσία, μια σχετική εταιρεία. Ε, οπότε θα με ενδιαφέρει να γνωρίζω τη γνώμη σας. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Χαίρομαι που είστε εδώ, γιατί έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα πριν από δύο χρόνια. Θέλω να τονίσω ότι δεν συμμερίζομαι τη γνώμη του Ντάνιελ Κασπάρη για το πώς ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Και στο σχέδιο του ψηφίσματος πιστεύω πως η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν βοηθά να βρούμε κάποιο κοινό σημείο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το σημείο 7 μάλιστα, στο σχέδιο αυτό. Ζητά από την Κομισιόν να προχωρήσει την διαβούλευση με τις αρχές της, ε, της Νορβηγίας ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε μια ικανοποιητική λύση για τα θέματα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε από κοινού για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η Νορβηγία είναι ένα κυρίαρχο κράτος μέσα στον ΕΟΧ και, και έχει κάθε δικαίωμα να έχει τους δικούς της κανόνες. Δεν υπόκειται στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Αλλά είναι γενικά καλό το ότι συνεχίζουμε να συζητούμε με το θέμα του, της Συμφωνίας Γενικευμένων Προτιμήσεων με τις Φιλιππίνες, όπου και πάλι εμπλέκεται το θέμα του άρθρου αυτού. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τις ε, ε, κυρώσεις που οποίες ανέφερε η κυρία Σάκη, να αντιμετωπίσουμε το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Πώς βλέπετε, πώς βλέπετε το γεγονός ότι δεν υπήρξε η παράδοση ορισμένων μορφών εξοπλισμού για την, ε, για την ζώνη από τους ε, Ρώσους. Μήπως αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο στο περιβάλλον Μήπως αυτό θα οδηγήσει σε δυσκολίες στην διερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου από την Καστρόμ και να αντιμετωπίσουμε μια οικολογική καταστροφή η οποία μπορεί να θίξει και την Ορβηγία. Θα ήθελα εδώ να έχω την άποψή σα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σχολιάσω αλλά σε επίπεδο ουσίας κυρία Σόλτς αναφέραστε στο ψήφισμα και όχι στο σχέδιο ψηφίσματος, γιατί υπήρξε αυτό το ψήφισμα του Ιουλίου 2013, απλώς για να έχουμε σαφήνεια σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Οι πράσινοι τώρα, εάν θέλουν να λάβουν το λόγο. Εάν όχι, ο κύριος ε, Γουλιέλμος Δαρτμούθιος. Τουλάχιστον στη δική μας επιτροπή υπάρχουν μερικοί που εκτιμούν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Νορβηγία είναι κυρίαρχη χώρα. Και φοβάμαι ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό όλοι μας οι συνάδελφοι σε άλλες, επιτροπέ. επιτροπές. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται για την διατήρηση του περιβάλλοντος ας πούμε πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα για τη διατήρηση των αποθεμάτων αλλιευμάτων στη Βόρεια Θάλασσα γιατί δεν είναι τμήμα της κοινή αλλιευτικής πολιτικής η Νορβηγία. Αλλιώς θυμάστε εκείνη την περίπτωση των ε, Ολλανδών αλλιέων που είχαν ε, πιάσει 25% των αλλιευμάτων της Βρετανίας. Τέλος πάντων. Έχω και ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τον πρεσβευτή. Η Νορβηγία είναι φυσικά μέλος της ΕΖΕΘ και ένα από τα χαρακτηριστικά της τελευταίας είναι ότι η ΕΖΕΣ ε, δέχεται και αυτή την ίδια ελευθερία κίνησης των ανθρώπων όπως η Ένωση. Η Ελβετία που είναι το άλλο θεμέλιο της ΕΖΕΣ έχει τελευταία ψηφίσει ότι δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία. Και το ερώτημα προς τον πρέσβη είναι, κάτε σας, πόσο ακόμα θα μπορέσει η Νορβηγία να, να, εφαρμόζει αυτή την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Μήπως θεωρείτε ότι η Νορβηγία πρόκειται να πάρει απαρόμοια στάση με της Ελιβετίας τα επόμενα πέντε χρόνια ας πούμε. Σας κατευχαριστώ. Έγινε ο πρώτος γύρος των πολιτικών ομάδων. Τώρα θα αρχίσει η συζήτηση για τους υπόλοιπους βουλευτάς μέλο, μέλη της Επιτροπής μας που μπορεί να θέλουν να κάνουν δηλώσεις ή σχόλια ή να θέσουν απορίες. Ορίστε εσείς παρακαλώ εκεί κάτω κύριε Μπένσον μου. Ευχαριστώ καταρχήν κύριε Πρέσβη για τα σχόλιά σας και για τη συνεργασία μας γενικότερα. Άκουσα ότι θέλετε να αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί για τα ψάρια και άλλα προϊόντα από τις θάλασσες, Αλλά η νέα κυβέρνηση δεν κατήργησε τους φόρους για ορισμένα τυριά, για το πρόβιο κρέας και λοιπά που ζητούσε η Ένωση. Εγώ νομίζω ότι αυτό παραβιάζει το άρθρο 19. 19. Αν θέλετε ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές μας, πρέπει να μας δώσετε το ίδιο δικαίωμα και για τις δικές σας αγορές και στη Γεωργία. Δεν θέλω να σχολιάσω πώς στηρίζετε τους αγρότες σας, κάντε ό,τι θέλετε γι' αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ίση πρόσβαση στις αγορές. Αυτό είναι το θέμα. Πρόσβαση στις αγορές. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως άλλος συνάδελφος θέλει να μιλήσει σε αυτή τη φάση, γιατί αν όχι, τότε λύγει και αυτός ο γύρος και στρεφόμαστε πάλι στον πρεσβευτή για να απαντήσει. Ακούσατε σχόλια, ακούσατε απορίες. Δεν είμαστε βέβαια στην Επιτροπή Αλληλείας αλλά Διεθνούς Ενυπορίου. Αλλά ανησυχούμε, ενδιαφερόμαστε και για τα θέματα των ηχθείων. Ορίστε κύριε πρέσβη μου. Ηχθείων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σημείωσα ότι δεν υπήρχαν πολύ φορούμενα ερωτήματα αλλά Τέλος πάντων, ήταν όλα πολύ πολύπλοκα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Γενικά, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οτιδήποτε λέτε και είπατε και μου μεταφέρατε, θα μεταφερθεί πιστά στις αρχές της κυβέρνησης και της χώρας μου. για τις διαφορές μας. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει τώρα, ξέρουμε ότι θα γίνει διαπραγμάτευση και συζήτηση και έχουμε και ένα πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις. Για μένα αυτό είναι πολύ ισχυρό και σταθερό πλαίσιο. Μέχρι τώρα βρίσκαμε πάντοτε λύσεις στις διαφορές μας και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. ε. Τώρα κατά πόσον οι πολιτικοί παίζουν με τη φωτιά ή όχι δεν το ξέρω. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλο και θα παραμείνω τέτοιος. Αλλά όπως σας είπα και πριν θα μεταφέρω το μήνυμά σας. Πλήρως μάλιστα. Αν μερικοί από, σας, μερικοί είπαν ότι δράσαμε με μη φιλικό τρόπο, εχθρικό τρόπο, αυτό δεν τον πιστεύω. Αλλά θα το μεταφέρω και αυτό. Και σας βεβαιώνω ότι δεν έχουμε παυλοφικά ανακλαστικά εχθρικά για σας. Δεν λέω ότι ποτέ δεν θα κάνουμε τίποτα που να το θεωρήσετε εχθρικό ή μη φιλικό, αλλά δεν είναι η πρόθεσή μας αυτή. Δεν το κάνουμε αυτόματα και επίτηδες. Γιατί είστε ο κύριος εταίρος μας εμπορικό. εμπορικός. Το ίδιο ισχύει και για το ότι έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι δεν κάνουμε διαβούλευση. Ότι δεν σας συμβουλευόμαστε. Δεν θέλω να διταχθώ σε απόψεις βουλευτών, αλλά ξέρω ότι και ο ίδιος έχω δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο σε διαβουλεύσεις ακριβώς και ο βαθμός της συνεργασίας μας απαιτεί να υπάρχει διαβούλευση. Ίσως σε ορισμένες συγκεκριμένε περιστάσεις να μην κάναμε αρκετή διαβούλευση. Αυτό ίσως, αυτό ίσως. Χαίρομαι γιατί τέθηκε το ερώτημα ενός βουλευτή που μας με ρώτησε πόσα πληρώνουμε. Δεν πληρώνουμε. Οι ΕΖΕΣ και η Νορβηγία αντιπροσωπεύουν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την τελευταία περίοδο και αυτό είναι μια συμβολή από την Νορβηγία μαζί με, την, με το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία για να συνεχίσει να υπάρχει οικονομική συνοχή. Αλλά δεν πληρώνουμε για την ΕΖΕΣ, δεν πληρώνουμε. Να, εδώ είναι το καταστατικό της ΕΖΕΣ. Και στόχος του ήταν να είναι όλοι ισότιμα μέλη να χορηγηθούν οικονομικά μέσα σε αυτή την πενταετή περίοδο, ε, όπως σας είπα, 1,8 δισεκατομμύρια για να μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Τώρα πώς οι εθνικοί νόμοι επηρεάζονται από αυτά τα 10.000 νομοθετήματα των τελευταίων 20 ετών στα πλαίσια της ΕΖΕΣ δεν το έχω υπολογίσει, ομολογώ, αλλά στην έκθεση που κάναμε πριν από ένα-δύο χρόνια, κάποιος από την κυβέρνηση υπολόγισε ότι ίσως 70%. Άλλοι λένε όμως όχι, όχι 70%. Αφού έχουμε το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο για τα κεφάλαιο, τις αγαθά και τους ανθρώπους, Δεν σημαίνει αυτό αυτόματα ότι αυξάνονται γεωμετρικά οι αριθμοί των νομοθετημάτων. Δεν έχω λοιπόν ακριβείς αριθμούς, αλλά σας ανέφερα περίπου αριθμούς που διάβασα κι εγώ και που νομίζω ότι απορρέουν από τα βασικά δεδομένα που ισχύουν για τη λειτουργία της ΕΖΕΣ. Πράγματι υπάρχουν πολλοί νόμοι και κανονισμοί που πρέπει να εφαρμόζονται. Ε, sanctions. Για τις κυρίσεις, κυρώσεις, συγγνώμη. Αυτό είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς τι σημαίνει. Γιατί είναι δύσκολο να ξέρει κανείς. Είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση αυτό το οποίο γνωρίζω πράγματι είναι το επίπεδο των εξαγωγών που έχουμε εμείς για τα αλληλευτικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που, επιβάλλει, που έχουμε επιβάλει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι σε ό,τι αφορά τον τομέα της προσφοράς που θα υπάρξουν επιπτώσεις. Δεν είναι όμως μια γραμμική εξέλιξη. Ξέρουμε ότι είναι πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν πρόκειται για επενδυτικά σχέδια, τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Δεν είμαι σε θέση λοιπόν να σας πω ότι το αποτέλεσμα έχει αυτό το μέγεθος. Όταν δούμε όμως τις κυρώσεις οι οποίες προέρχονται από τις συμφωνίες μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι μόνο οι κυρώσεις, θα είναι το γενικό επενδυτικό κλίμα το οποίο θα επηρεαστεί και μόνο σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο θα μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των κυρώσεων και θα μπορέσουμε να ξέρουμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι προσπάθησα έτσι εν μέρη να απαντήσω το ερώτημα για το περιβάλλον. Όλα αυτά που κάνουμε στον ακραίο βορρά έχουν γίνει στην αντιμετώπιση της εξόρυξης πετρελαίου μέσα σε πάρα πολύ αυστηρά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό εξαρτάται από το τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν οι Ρώσοι. Σας ευχαριστώ πάντως για όλα αυτά που μας έχετε πει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα προκύψει σε μια περιοχή η οποία είναι κέρια στρατηγικά για μας και θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρούνται τα πιο αυστηρά πρότυπα για το περιβάλλον στην αρχική ζώνη. Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και η ΕΖΕΣ. Ναι, μέσα στην ΕΖΕΣ βρίσκεται η Νορβηγία. Ενώ έχει διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συρρυκνωθεί η ΕΖΕΣ. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να ήμουν στη γραμματεία της ΕΖΕΣ στη Γενέβη. Τότε ήταν Πολύ σημαντική η ΕΖΕΣ. Δεν υπάρχει τώρα τίποτα στην Ορβηγία που να δίνει την εντύπωση ότι εμείς θα φερθούμε πως η Ελβετία. Κάθε άλλο εμείς έχουμε τονίσει πάντα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι ένα πάρα πολύ κέριο στοιχείο της ενιαίας αγοράς. μέσα στην οποία είμαστε ενσωματωμένοι με τη συμφωνία του ΕΟΧ. Για τα αλλιεύματα έθιξα αυτό το θέμα γιατί είναι πραγματικότητα. Θέλουμε να βελτιώσουμε την αγορά μας για τα προϊόντα αυτά. ο καθένας πρέπει να κοιτάξει και τα δικά του συμφέροντα σε αυτήν την περιοχή. Όταν όμως ξαναγυρίζω στο θέμα που τέθηκε στην αρχή της συζήτησης, ξέρω ότι έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ληφθεί αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γεωγραφική ένδειξη προέλευσης. Όταν λοιπόν προσπαθώ να δημιουργήσω μια γενική εικόνα να σας παρουσιάσω, προτιμώ <clears throat> πάντα να τονίζω και αυτό, ότι έχουμε μια πραγματική πλατφόρμα μέσα στην οποία μπορούμε να βρούμε τη λύση των προβλημάτων. Και θέλω να σας ευχαριστήσω με αυτή την τελευταία αισιόδοξη σκέψη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ και μας δώσατε ε, τις πληροφορίες όλες αυτές. Φυσικά το εμπόριο σημαίνει διαπραγματεύσεις, αλλά για αυτήν εδώ την Επιτροπή μας ε, σημαίνει και εκτεταμένες αρμοδιότητες ε, συμπεριλαμβανομένες της παρακολούθησης των συμφωνιών. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι για τις διάφορες διαδικασίες και την παρακολούθηση αυτών των διαπραγματεύσεων και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις σχέσεις μας τις εμπορικές. Ευχαριστώ πολύ εξοχότατε. And, uh, uh, now, uh, colleagues, the next... Και τώρα, συνάδελφοι, το επόμενο σημείο είναι, μάλλον τα δύο επόμενα σημεία είναι η κοινή συζήτηση, σημεία 12 και 13, για δύο προτάσεις για κωδικοποίηση ισχυωσών νομοθεσιών, κοινών ε, κανόνων της Ένωσης για ε, την ε, μέτρα εποπτείας των εισαγωγών. Οι προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν ουσιαστικές αλλαγές και ε, παρουσιάζονται υπό τη μορφή δύο αναθεωρήσεων μιας διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητά μας να τροποποιήσουμε τις προτάσεις. Έχουμε το σημείο 12, την εισαγωγή προϊόντων υφαντουργίας που δεν καλύπτονται από άλλες συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους κανόνες της Ένωσης. Ε, και το σημείο 13 είναι εισαγωγέ εισαγωγές από συγκεκριμένες τρίτες, από ορισμένες μάλλον τρίτες χώρες. Και εδώ έχουμε recast. Καλό λοιπόν τον κύριο Λουίτζι Τσιμάλια, τμήματάρχη, τμήματάρχη της ε, μονάδας ε, που είναι αρμόδια για το Διεθνές Εμπόριο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη εισήγηση σε σχέση με την χρήση των νομοθετικών τεχνικών κωδικοποίησης και ε, αναθεώρησης. Και βεβαίως η Κομισιόν είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορά αυτό το θέμα. Υπάρχουν δύο νομοθετικές ε, τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως ε, με στόχο την απλοποίηση υφιστάμενων νομοθεσιών. Οι κανόνες που αφορούν την συγκεκριμένη χρήση αυτών των δύο νομοθετικών τεχνικών καταγράφονται σε δύο διαφορετικές ε, διοργανικές συμφωνίες. Μία αφορά την κωδικοποίηση και η άλλη την αναθεώρηση, η RICAST. Θα ήθελα να σας παραθέσω δύο αρκετά σημαντικά ε, σημεία των δύο διοργανικών συμφωνιών Το πρώτο αφορά την ορισμό του τι είναι κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση σημαίνει την διαδικασία για την ε, κύρωση πράξεων που πρόκειται να κωδικοποιηθούν και την αντικατάστασή τους από μία μόνο πράξη που δεν περιέχει ουσιαστικές αλλαγές αυτές τις πράξεις. Όπως βλέπετε λοιπόν από αυτό το πρώτο σημείο της συμφωνίας, το διακριτικό χαρακτηριστικό μιας κωδικοποίησης είναι η πλήρης απουσία οποιονδήποτε ουσιαστικών αλλαγών σε σχέση με την υφιστάμενη ισχύουσα μάλλον νομοθεσία. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έννοια όσον αφορά την κωδικοποίηση και επαναλαμβάνεται ε, και σε άλλα σημεία της διοργανικής συμφωνίας, ε, δηλαδή το σημείο 3 που λέει ότι η Κομισιόν δεν θα συμπεριλάβει στις προτάσεις κωδικοποίησης ουσιαστικές αλλαγές στις πράξεις που πρέπει να κωδικοποιηθούν. Και το σημείο 6 της ίδιας συμφωνίας ε, λέει ότι στόχος της πρότασης της Κομισιόν, δηλαδή η ορθή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, αποτελεί την, ε, ε, ε, ε, την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή από πλευρά του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου. Σημαντικό επίσης είναι στην διαδικασία κωδικοποίησης ότι η φυσιολογική νομοθετική διαδικασία της Ένωσης θα πρέπει να τηρηθεί πλήρως. Τώρα, σε σχέση με την κωδικοποίηση όπου οι ουσιαστικές αλλαγές λείπουν τελείως. Το recast, η αναδιατύπωση, σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν και κάποιες ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με ένα υφιστάμενο νομικό κείμενο. Και πάλι θα ήθελα να παραθέσω από το σημείο της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την αναδιατύπωση όπου μπορείτε να βρείτε και ορισμό της ε, ε, αναδιατύπωσης, η recast, Πρόκειται δηλαδή για την υιοθέτηση μιας νέας νομοθετικής πράξης που ενσωματώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τις ουσιαστικές αλλαγές, τροποποιήσεις που γίνονται μέσω μιας προηγούμενης πράξης και καθώς και τις μη τροποποιημένες διατάξεις της ίδιας πράξης. Και πάλι, όπως και για την κωδικοποίηση, η νέα νομική πράξη αντικαθιστά και ακυρώνει την προηγούμενη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν στην, ε, και εδώ θα πρέπει να ακολουθηθεί πλήρως η φυσιολογική νομοθετική διαδικασία που ισχύει στην Ένωση. Πολύ σύντομη λοιπόν παρουσίαση όσον αφορά τις δύο αυτές τεχνικές κωδικοποίησης και αναδιατύπωσης. Αλλά βεβαίως, εάν υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, είμαστε στη διάθεσή σας. Τώρα, όσον αφορά τις δύο προτάσεις αναδιατύπωσης που έχει υποβάλει το περισμένο καλοκαίρι η Κομισιόν. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο του αποκαλούμενου Trade Omnibus. Στις αρχές ε, του τρέχοντος έτους δύο κανονισμοί, ο υπαριθμών 37 και 38 του 2014, υιοθετήθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα. Όταν, οι δύο αυτοί, όταν εγκρίθηκαν αυτοί οι δύο κανονισμοί, η Κομισιόν δεσμεύτηκε να κωδικοποιήσει τις πράξεις που ε, τροποποιούνταν μέσω αυτών των δύο κανονισμών. Το σύνολο των πράξεων που τροποποιήθηκαν από τους κανονισμούς 37 και 38 θα πρέπει να είναι 36 αν δεν κάνω λάθος. Οι περισσότερες από αυτές τις πράξεις υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν μέσω προτάσεων κωδικοποίησης ή αναδιατύπωσης. Οι περισσότερες αυτές πράξεις απλώς έχουν κωδικοποιηθεί, ενώ κάποιες από αυτές τις πράξεις, από ό,τι φάνηκε, χρειάζονταν να γίνουν κάποιες ελαφρές αλλά ουσιαστικές τροποποίησεις. Γι' αυτό ακριβώς οι δύο προτάσεις που σας έχουν υποβληθεί σήμερα έχουν ε, υποβληθεί υπό τη μορφή recast, δηλαδή αναδιατύπωσης. Γιατί δεν περιλαμβάνουν απλά μόνο κωδικοποίηση των ισιών των κανόνων που περιλαμβάνονται στους δύο κανονισμούς, αλλά και κάποιες μικρές ε, αλλαγές. Υπάρχουν ε, βέβαια και μεμοράντα, υπομνήματα μαζί που συνοδεύουν αυτές τις ε, προτάσεις και λένε ότι ξεκίνησε η διαδικασία κωδικοποίησης αρχικά αλλά κατέστη αναγκαίο να γίνουν κάποιες τροποποίησεις και άρα μετετράπησε διαδικασία αναδιατύπωσης. Οι αλλαγέ αυτές πάντως ε, θεωρώ ότι μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι πολύ απλές ελαφριές αλλά ουσιαστικές και είναι αυτές που συνήθως ε, θεωρούμε ότι είναι απλά τεχνικής φύσης ε, πρέπει να υπογραφούν και άρα να θεωρήσουμε ε, Ε, λοιπόν ότι πρόκειται για ε, κωδικοποίηση με κάποιες μικρές ε, τροποποίησεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Όντως, αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ασχολείται με τη διαδικασία αναδιατύπωσης. Και μετά από αυτή την πρώτη παρουσίαση από την πλευρά της Κομισιόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, ο Γιάρος Λαβόας από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Βαλές. Εγώ ζήτησα να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή απόψε για το θέμα αυτό, προτού παρουσιάσω το σχέδιο εκθεσή μου, για να έχω μια καλύτερη αίσθηση για το τι θέλουν οι πολιτικές ομάδες να κάνουμε για αυτό το θέμα. Οι δύο αυτές προτάσεις θα κωδικοποιήσουν, θα κωδικοποιήσουν τους τωρινούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τροποποιηθεί πολλές φορές και επομένως η παγιοποίησή τους τους κάνει πιο φιλικούς προς τον χρήστη. Οι προτάσεις αυτές όμως περιλαμβάνουν κάποιες ουσιαστικές τροποποίησεις. Η Κομισιόν της παρουσιάζει ως μία αναδιατύπωση της νομοθεσίας και όπως, όπως λέτε κύριε Πρόεδρε, περιορίζεται η δυνατότητά μας ως συνομοθέτου να τροποποιήσουμε αυτές τις προτάσεις. Οι ουσιαστικές αυτές αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν ε, εμφανίζονται με φαιά στοιχεία σε αυτή την πρόταση. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή μας αντιμετωπίσει μια αναδιατύπωση μιας ε, νομοθετικής πρότασης ως αρμόδια επί της Επιτροπή. Να σας εξηγήσω λοιπόν πώς έχει η διαδικασία. Είναι φυσιολογική νομοθετική διαδικασία με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που εφαρμόζονται σε σχέση με τις τροπολογίες. Καταρχήν, οι τροπολογίες αυτές είναι παραδεκτές για αυτό το κείμενο το οποίο είναι φαίο, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να τροποποιηθούν τα μη φαιά τμήματα της πρότασης, αλλά με την ε, προϋπόθεση ότι θα πρέπει αμέσως να αναφέρουμε την πρόθεσή μας να κάνουμε κάτι τέτοιο προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Μια άλλη ιδιαιτερότητα στη διαδικασία αναδιατύπωσης θα πρέπει να είναι ο έλεγχος από την πλευρά των τριών θεσμικών οργάνων, Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και, και ο έλεγχος από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες των τριών αυτών φορέων και από την Επιτροπή η Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν κατά πόσο η Κομισιόν έχει περιοριστεί στο να κάνει αυτές τις τροπολογίες οι οποίες ε, μπορούν να εντοπιστούν από το φαιό κείμενο. Και η νομική υπηρεσία όταν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο μπορεί να τα δώσει τα στοιχεία αυτά στη νομική επιτροπή και η νομική επιτροπή κάνει και αυτή τον έλεγχο τον αντίστοιχο. με έχουν πληροφορήσει ότι την επόμενη εβδομάδα θα εγκρίνει τη γνωμοδότηση της Νομική Επιτροπή και ξέρω ότι και από την πλευρά των κατών μελών η προθεσή του είναι να συμφωνήσουν με την πρόταση τη Κομισιόν ως έχει. Εν τέλει θα ήθελα να πω ότι οι προτάσει αυτέ συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο νομοθετημάτων <clears throat> που έπρεπε να ε, ενσωματωθούν στο νέο πλαίσιο των εξουσιοδόση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων ήταν τμήματα του Omnibus, του νομοθετήματος Omnibus 1 και αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Σε ό,τι τώρα αφορά την ουσία των προτάσεων, τα θεά τμήματα, έχουμε κάποιες τεχνικές προσαρμογές, ε, διορθώσεις φαλμάτων τα οποία έχουν διαπιστωθεί και στον γενικό κανονισμό ο οποίος καλύπτει τις εισαγωγές που δεν είναι κλωστοφαντουργικά αγαθά και αφαιρούνται με χώρες όπως η Ρωσία, η Αρμενία, τα Τζικιστάν και η Βιετνάμ από το παράρτημα γιατί τώρα έχουν γίνει μέλη του ΠΟΕ και αυτό σημαίνει ότι η κάλυψη της πρότασης περιορίζεται στο Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, τη Λευκορωσία, τη Βόρεια Κορέα, Τουρκμενιστάν αλλά και Ουσμπεκιστάν. Και τέλος, ό,τι αφορά την πρόταση για τις εισαγωγές κλώστα εφαντουργικών, η προτέρα διαδικασία λήψης απόφασης στο άρθρο 23 έχει αντικατασταθεί από μια διαδικασία απόφασης η οποία έχει τύχει απόφαση στο νομοθέτημα Omnibus 1. Όπως ξέρετε, ο τομέας των κλωστοφαντουρικών είναι πολύ ευαίσθητος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι μόνες χώρες από τις οποίες εισάγει κλωστοφαντουργικά προϊόντα η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλες διευθετήσεις ή από άλλες κανόνες εισαγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το GPA, το GSP και το EBA είναι η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα. Ο κανονισμός θεσπίζει ετήσια ποσοτικά όρια για ένα αριθμό κλωστοφαντουργικών προϊόντων από τις χώρες αυτές και επιτρέπει το να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ο κανονισμός επιτρέπει την παρακολούθηση και την εποπτεία και τα μέτρα διαφύλαξης όταν οι εισαγωγές κλωστοφαντουργικών ξεκινούν από άλλες, από τρίτες χώρες και μπορεί να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα προς τους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να πω τώρα και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να ακούσω τα δικά σας σχόλια και προτάσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. And uh, now, uh... Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Σκιώδης. Από τους Σοσιαλιστάς η Αλήσια Μόσκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την ε, πολύ λεπτομερή εισήγηση από τεχνικής αλλά ε, αλλά και από άποψη περιεχομένου. Η θέση μας αυτή τη στιγμή ε, είναι θέση στήριξης στη αίτημα της ε, Κομισιόν για αναδιατύπωση ε, και Πιστεύουμε πως αυτό θα απλοποιήσει και θα ενημερώσει ολόκληρη την νομοθεσία. Πρόκειται δε για, βασικά για τεχνικές, ε, τεχνικά θέματα. Δεν έχουμε αντίρρηση λοιπόν γιατί πρόκειται στην ουσία για διορθώσεις ε, όσον αφορά την ενημέρωση αλλά και την συνέπεια των, με τις διαπραγματεύσεις μας, όπως αυτές προχώρησαν ε, με κάποιες χώρες. Χρειαζόταν λοιπόν μια ενημέρωση και άρα και επί της ουσίας θεωρούμε πως μπορεί να εγκριθεί αυτή η πρόταση. Περιμένουμε λοιπόν να μας δοθεί και η απάντηση από την νομική μας υπηρεσία, ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much for the, uh, the conservatives. Mrs. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακλάρκιν από τους συντηρητικούς. To us. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκιώδης εισηγητής. So, if it's, uh, if it's not the case, then for... Uh... Εάν δεν είναι κάποιος εδώ, η κυρία Σάκη από την άλλη. Thank you, Chair. Uh, I'll also be very... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα είμαι σύντομη. Όλα αυτά είναι πολύ τεχνικά αλλά χαιρετίζουμε την πρόταση αναδιατύπωσης γιατί είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία να είναι διαφανής και εύληπτη. Χαιρόμαστε επίσης για την αλλαγή στο άρθρο 23 που δίνει τη δυνατότητα στην παράταση ορισμένων αδειοδοτήσεων εισαγωγών για να διευκολυνθεί το εμπόριο και να μειωθεί η γραφειοκρατία. Προς στιγμήν δεν προσκοπεύουμε να καταθέσουμε καμία τροπολογία. Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στους συντηρητικούς. Κύριε Λούνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι καινούριο βουλευτής στο Κοινοβούλιο και μόλις έμαθα τι σημαίνει κοινή συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν για το λόγο. Και φυσικά θα συνεργαστώ με όλους και όλες σας τα επόμενα χρόνια και ελπίζω να είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για τη συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται βέβαια ιδιαίτερα τεχνική. Καλό είναι να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε ακριβώ τα τεχνικά για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και επίσης, ίσως επειδή είμαι καινούριο, έχω ορισμένες πρακτικές απορίες. Από τη μία δηλαδή. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν για ποια προϊόντα μιλάμε, για ποια διαπραγματευόμαστε. Ποια είναι τα προϊόντα που ανταλλάσσουμε με τις χώρες αυτές. Ποιο είναι το ύψος του εμπορίου μας, ας πούμε με την Νότια Κορέα. Δεν νομίζω ότι εξάγουμε υφάσματα, αλλά τι ακριβώς εξάγουμε και τι εισάγουμε. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας απαντήσει δεύτερον. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό μήπως μπορούμε να, μπορεί να γίνει μια επισκόπηση. Τα τελευταία χρόνια μερικά κράτη-μέλη ζήτησαν επιτήρηση μέτρα εποπτείας. Υπάρχουν τίποτε στοιχεία περί αυτού. Έχει γίνει αυτή η επιτήρηση ή η εποπτεία. Ευχαριστώ πολύ. Την κούε τώρα. Δεν βλέπω όμω εδώ τον κύριο Σόλτς. Η πράσινη λοιπόν. Πράσινη. Δυστυχώς δεν είναι ο εισηγητής μας ο Σκιώδης εδώ παρόν, αλλά για μένα έχουν λεχθεί τα σημαντικότερα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε για ποιον όγκο εμπορίου μιλάμε αυτή τη στιγμή. Uh, thank you very much. I go now. Σας ευχαριστώ. Η ομάδα του EFTD δεν θέλετε να πείτε τίποτα. Ωραία. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους μας αν κάποιος άλλος βουλευτής θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν φαίνεται να θέλει κανείς. Εάν όχι, στρέφομαι και πάλι προς την Κομισιόν, διέφθηκαν ορισμένα ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν και θέλουμε να δούμε αν η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Σας ξαναδίνω λοιπόν τον λόγο. δεν είναι καλή μέρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνεται σε ό,τι αφορά την παροχή απαντήσεων. Γιατί και το πρωί τα ίδια προβλήματα είχαμε. Σας ξαναρωτάω, μήπως είναι κανείς διαθέσιμος να απαντήσει τα ερωτήματα που έχουν θέσει τα μέλη του Κοινοβουλίου. Εάν όχι, και αυτό είναι λίγο προβληματικό. Okay, uh, Θα πρέπει να ξαναγυρίσω λοιπόν στον εισηγητή μας, τον κύριο ο, οποίος ε, έχει το λόγο για να κάνει τις καταληκτικές του παρατήρησεις. Κύριε Μία από τις προτάσεις βέβαια έχει να κάνει με τα κλωστοεφαντουργικά προϊόντα. ο λόγο που ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό ήταν για να έχω κάποια ιδέα για τι ουσιαστικέ πρώτα στην πρόταση. Εμεί όλοι συμφωνούμε όμως ότι αυτό το οποίο προήλθε από την πρόταση της Κομισιόν είναι θετικό και επομένω να το αφήσουμε όπω είναι. Αυτό είναι ίσω το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση και στην στα έδρα τη Κομισιόν. Αν θέλει κάποιο λοιπόν να λάβει το λόγο, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Μαριάννα Ιγνατέσκου από την ε, νομική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και συντονίζω τις ε, προτάσεις αλλαγής και αναδιατύπωσης. Έχω δύο ερωτήματα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να έχετε μια συνολική εικόνα για τα μέτρα εποπτείας βάσει του κανονισμού για τα κλωστοϊφαντουργικά ή του κανονισμού για τις διαφυλάξεις. Αυτά είναι θέματα ουσίας, δεν είμαστε έτοιμοι όμως να απαντήσουμε. Αλλά αν χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να σας διαβιβάσουμε αργότερα. Ευχαριστώ. Εντάξει. Κάντε λοιπόν τις απαραίτητες επαφές γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να έχουν αυτές τις πληροφορίες. Και μου λέει η γραμματεία ότι θα θέλαμε να ξέρουμε και αν το Συμβούλιο έχει κάποια σχέδια για αυτές τις διαδικασίες ε, αναδιατύπωσης αν θέλει να προτείνει κάποιες ε, προτάσεις τροποποίησης. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο λοιπόν έχει κάποια σχόλια που θέλει να κάνει. Δεν φαίνεται ότι το Συμβούλιο θέλει να κάνει κάτι και πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογό μας και τα επόμενα βήματα η Κομισιόν όμως Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πληροφορίες σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου. Είχαμε μια συναντρίαση της ομάδος εργασίας του Συμβουλίου για την νομοθετική κωδικοποίηση όπου Εγκρίθηκαν όλες τις προτάσεις κωδικοποίησης και επίσης είχαμε κάποιες συναντήσεις της ομάδος εργασίας που είναι αρμόδια για το διεθνές εμπόριο όπου έγιναν και σημαντικές πρόοδοι για τα θέματα αυτά και όπου εάν δεν απατώμε υπήρξε κάποιος ήδη βαθμός συμφωνίας που επετεύχθη. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να προκύψει μια συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου αρκετά σύντομα, τουλάχιστον σε επίπεδο ομάδος εργασίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Today indeed seems to be a difficult day for, uh, for our inter... Στα δύσκολα βρίσκεται η διαθεσμική συνεργασία, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσω αυτό το σημείο και να έρθω στα επόμενα βήματα βάσει του προσωρινού χρονοδιαγράμματος που συνέταξε ο εισηγητής. Η, τοσία σχέδιο θα αντιμετωπιστεί στην εδρία στη ΣΥΝΤΑ τον Δεκέμβριο 3 και 4. Η ψηφοφορία μας βέβαια, η ημερομηνία ψηφοφορίας θα εξαρτηθεί από την γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής και αν γίνει αυτό στις 3 και 4 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε το σχέδιο αυτό και θα έχουμε μια προθεσμία τροπολογιών μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία στις 21 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο του 2015 εάν θέλει ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ και πέραμε στο επόμενο σημείο το σημείο υπαριθμών 14 είναι ο κατεξουσιοδότης κανονισμός για την τροποποίηση του άρθρου 3 στον κανονισμό 978-2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με ένα σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων πρόκειται για τις Φιλιππίνες και υπό μορφή εισαγωγικής παρατήρησης. Σας υπενθυμίσω στις 19 Αύγουστου του 2014 η Κομισιόν ενέκρινε μια κατεξουσιοδότηση πράξη που προτείνει να δοθεί καθεστώς GSP συν στις Φιλιππίνες. Αυτή η ειδική λοιπόν ε, ρύθμιση είναι ένα κίνητο για αηφόρο αντιμετώπιση και καλή διακυβέρνηση και δίνει δεσμολογικές προτιμήσεις σε ευάλωτες χώρες οι οποίε εφαρμόζουν 27 κέρδιες συμβάσει. τελευταία μεταρρύθμιση του κανονισμού GSPC επέτρεψε στι Φιλιππίνες να ζητήσουν το κατεστώς GSPC που έγινε πραγματικότητα η πρόταση αυτή το Φεβρουάριο. Αν γίνει δεκτή η αίτηση των Φιλιππινών θα είναι 14η χώρα η οποία θα ενταχθεί στο σύστημα GSP-SYN. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουν δύο μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο μήνες να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Έτσι, ε των διαφόρων πολιτικών ομάδων, ομάδων οι συντονιστές των ε, πολιτικών ομάδων μου ζήτησαν να υπάρξει μια αναβολή ως το Δεκέμβριο, ώστε να μπορέσουν τα μέλη της Επιτροπής μας να έχουν μια καλά εμπεριστατωμένη άποψη. Έχουμε τώρα μια ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν και τον Πρεσβευτή των Φίλιππινών που θέλω να χαιρετήσω στην αίθουσά μας, ώστε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να είναι πλήρως πληροφορημένα και να αξιολογήσουν την κατάσταση. Ο κ. Αλέν Καντέκ είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα λάβει και αυτό το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Μετά τη συζήτηση τα, μέτρα, τα μέλη της ΙΝΤΑ θα έχουν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου για να προτείνουν μια αντίρρηση στην κατεξουσιοδότηση πράξη που δίνει στις Φιλιππίνες το καθεστώς του GSP συν. Και δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes, thank you, Chairman. Μάλιστα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε το γενικεμένο σύστημα προτιμήσεων συν. Θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω ότι τα μέλη που ίσως δεν γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το εργαλείο όπως ξέρουμε είναι ένα εργαλείο γενικευμένων κινήτρων για καλύτερη διακυβέρνηση και που χορηγείται με βάση αίτηση εθελοντικά σε χώρες που θέλουν να αναλάβουν ορισμένες πρόσθετες δεσμεύσεις για την εφαρμογή 27 διεθνών συμβάσεων που καλύπτουν μεγάλο φάσμα θεμάτων, πολέμηση διαφθοράς κλπ. κλπ. Όπως σας είπα λοιπόν είναι κίνητρα, είναι συλλογή κινήτρων ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να βοηθηθούν να εφαρμόσουν πραγματικά αυτές τις ε, ρήτρε δεν έχει στόχο να καταλήξει σε τέλεια εφαρμογή όλων των ενδιαφερμένων χωρών, αλλιώς θα έπρεπε να καλύπτει και την Ελβετία και την Νορβηγία και άλλες χώρες, όχι μόνο αυτές. Τα κριτήρια που θεσπίζει για τις χώρες που θέλουν να πάρουν να κάνουν αυτό το βήμα είναι απλά. Και τα εφαρμόζουμε, τα εφαρμόζαμε μέχρι, τα εφαρμόσαμε σε 13 περιπτώσεις που τις έχουμε συζητήσει πέρυσι εδώ στην Επιτροπή μας για τις 13 χώρες που είναι ήδη μέλη του συστήματος αυτού GSP+. Υπενθυμίζω βέβαια ότι πρέπει τα κριτήρια αυτά να εφαρμόζονται με αντικειμενικό και ισότιμο τρόπο και φυσικά συνεπώς. Οι Φιλιππίνες έκαναν, υπέβαλαν ένα τέτοιο αίτημα φέτος, το εξέτασε η Κομισιόν και είδε ότι πληρεί τα κριτήρια. Και στις 9 Αυγούστου αποφασίσαμε να προτείνουμε οι Φιλιππίνες να ενταχθούν στο σύστημα GSP+. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια αυτά. Πρώτον που είναι και το μόνο οικονομικό κριτήριο είναι κατά πόσον υπάρχει κάποια ευαισθησία ως προς τις εισαγωγές προς την Ένωση. Δεύτερο κριτήριο η έγκριση και κύρωση των 27 αυτών συμβάσεων και εξετάζουμε βέβαια και τα συμπεράσματα των εποπτικών σωμάτων για την εφαρμογή αυτών των συμβάσεων γιατί υπάρχει, η κάθε μία έχει ένα διεθνές σώμα που τις εποπτεύει. Δεν πρέπει λοιπόν στα συμπεράσματα αυτά να λέει ότι υπήρξε σοβαρή έλλειψη στην εφαρμογή των συμβάσεων ούτε να έχει λάβει η χώρα μέτρα που να ακυρώνουν καμία από τις ρήτρες τους. Και φυσικά πρόκειται για κοινή επιχείρηση και δέσμευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σχετίζεται άμεσα με αυτό που θα κάνουμε μόλις μπει μια χώρα στο σύστημα GSP+. Σύμφωνα με την τελευταία της μεταρρύθμιση, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μας δίνουν την εντολή να επιτηρήσουμε στενά τις χώρες αυτές για να δούμε πώς εφαρμόζουν τις 27 συμβάσεις. Πρέπει να αναλάβουν δέσμευση, να συνεργαστούν μαζί μας και με τους διεθνείς οργανισμούς που εφαρμόζουν τις συμβάσεις, να δεχτούν επιτήρηση και φυσικά να μας χορηγήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την αξιολόγηση της κατάστασης. Και την αξιολόγηση αυτή τη χρειαζόμαστε γιατί όπως ξέρετε πρέπει τελικά να σας υποβάλουμε και σε εσάς και στο Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια μία έκθεση. Η επόμενη θα είναι του χρόνου για το πώς εφαρμόζουν τις συμβάσεις οι χώρες, οι ενταγμένες χώρες. Πέρυσι δημιουργήθηκε ένα σύστημα εποπτείας που βασίζεται σε δύο θεμέλια. Το πρώτο είναι ένας κατάλογος θεμάτων που τον λέμε scorecard που συμπεριλαμβάνει όλες τις ελλείψεις που έχουν σημειωθεί στην εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και που έχουν παρατηρήσει αυτές οι ενδιαφερόμενες χώρες. Τις ελλείψεις αυτές τις αναφέρουμε στους ενδιαφερόμενους και περιμένουμε απάντηση για το πώς θα τις αντιμετωπίσουν. Δεύτερον είναι ο διάλογος GSP+, δηλαδή. Δεν περιοριζόμαστε δεν, να περιμένουμε απαντήσεις, αλλά χρησιμοποιούμε ό,τι κανάλι διαθέτουμε, ε, εμπορικές επιτροπές, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 13 χώρες που είναι ενταγμένες στο σύστημα αυτό στο Πακιστάν, Γουατεμάλα, το Περού, Γεωργία, Αρμενία κλπ. κλπ. Το έχουμε κάνει αυτό. Το καινούριο θέμα στη μεταρρύθμιση του συστήματος δεν είναι τόσο τα κριτήρια ένταξης που όπως σας είπα είναι απλά, αλλά η εποπτεία ακριβώς αυτή της εφαρμογής του συστήματος και των συμβάσεων από τις χώρες αυτές και η εφαρμογή των δεσμεύσεων που μας έχουν δώσει την αξιολόγηση την κάνουμε και μέσα στο χρόνο δηλαδή. Μερικά από τα έγγραφά μας όπως τα scorecards που σας έλεγα δείχνουν ότι υπάρχει μακρύς κατάλογος ελλείψεων ή θεμάτων που καμιά φορά είναι λίγο ενοχλητικά στην ανάγνωση αλλά δεν αναμένουμε καμία ξαφνική ή μαγική λύση μέσα σε μια μέρα ή δύο μήνες. Γίνεται προσπάθεια να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να προχωρήσουν και μέσα στο χρόνο. Εν τω μεταξύ βέβαια το τρίτο θεμέλιο της εποπτείας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών που κάνουμε μεταξύ χωρών μελών και με την Επιτροπή σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μια νέα θεματική ομάδα που έχει δημιουργηθεί το, η ομάδα εποπτείας του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. σταματώ εδώ, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι στο τέλος της συζήτησης. Εδώ δώστε μου τρία λεπτά παραπάνω για να αναφέρω κάτι που σχετίζεται με το σύστημα αυτό και αφορά την ένταξη της Κένιας στο σύστημα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές ως προς την κατεξουσιοδότηση πράξη για την ένταξη της Κενίας. Τώρα όμως συνεχίζει ο διάλογος για τις Φιλιππίνες και έχουμε τον πρέσβη των Φιλιππινών εδώ σήμερα, την κυρία Βικτόρια Μπατακλάν, την οποία χαιρετίζω. Εξοχοτάτη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τους βουλευτές που μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις σκέψεις μας επ' αυτού. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Ήθελα να πω ότι δεν έχω τίποτα να προσθέσω, αλλά χαιρόμαστε για αυτή τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να χορηγήσουμε μερικές πληροφορίες που έχουν πολλές φορές ζητηθεί επίσημα από τους βουλευτές. Να σας πω και κάτι προσωπικό. Εγώ όλη μου την καριέρα με το GSP ασχολήθηκα στη Γενέβη παλαιότερα και δεν είχα καταλάβει ότι θα τελείωνα την καριέρα μου πάλι με το ίδιο θέμα. Πάλι για το GSP. Τώρα όμως είναι το GSP συν και όταν το πρωτοάκουσα και τα κριτήρια και αυτά είπα α, άλλαξαν τα πράγματα. Παλιότερα οι προτιμήσεις ήταν ανεφόρων και θεωρούνταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του διαλόγου Αλλά άλλαξαν τα πράγματα με το χρόνο και η απλοποίηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιτήρησή τους, η υποπτία τους, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος έχουν γίνει πια μόνιμο τμήμα όλων μας των σχέσεων και δραστηριοτήτων. Αυτό δεν μας πειράζει, το χαιρετίζουμε. Ζητήσαμε όντως να μπούμε στο σύστημα GSP+, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είμαστε γνώμονες που η Κομισιόν και το Συμβούλιο τους τελευταίους δύο μήνες θεώρησαν την αίτησή μας ε, σωστή και είμαι σίγουρη ότι με τις ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών θα μας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο και οι βουλευτές εγκρίνοντας και αυτή την ένταξή μας. Το GSP Plus είναι πολύ σημαντικό για τις Φιλιππίνες το χρειαζόμαστε πράγματι. Έχουμε ωφεληθεί από το παλιό GSP και από χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά είμαστε χώρα που χρειάζεται ακόμα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της, να κερδίσει περισσότερα, να κάνει περισσότερες επενδύσεις, να είναι πιο ανταγωνιστική, διότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για την παγκόσμια ανάπτυξη ακόμα δεν έχει λυθεί για μας. Και γι' αυτό προσβλέπουμε πάρα πολύ στο GSP Plus για τους παραγωγούς μας, για τους μεταποιητές μας, για τους βιομηχάνους μας, για τους αλληλείς μας και για όλους τους τομείς που θα ωφεληθούν. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι επιπτώσεις του συστήματος θα επηρεάσουν τη ζωή πολλών στις Φιλιππίνες που ζουν στην Ήπεθρο και όπου σημειώνονται μεγάλα ποσοστά ανέχειας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά τα καινούργια κριτήρια ή κίνητρα όπως λέγονται τώρα θα έχουν θετικό αποτέλεσμα στη ζωή των κατοίκων των Φιλιππίνων. Όπως είπε και ο Νορβηγός συνάδελφος προηγουμένως, για να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά, έχουμε 50 χρόνια σχέσεις οι Φιλιππίνες με την Ένωση και γι' αυτό και ο πρόεδρος μας τον περασμένο μήνα ήρθε εδώ να επισκεφθεί τα όργανα και συζητήθηκαν και πάλι γενικότερα τα θέματα των διμερών μας σχέσεων. Η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής μας και εμπορικός μας εταίρος και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ σε θέματα και ασφαλείας και πολιτικά ως προς την διαδικασία ειρήνευσης ας πούμε στις Φιλιππίνες. Για πράγματα το οποίο είμαστε δύο για να επικεντρωθώ τώρα ειδικά στο GSP+, Plus ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και παρεμφερή θέματα, όχι αποκλειστικά για τα κριτήρια, τα οποία δεχτήκατε, αλλά στη συζήτησή μου με πολλούς από εσά ε, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, μπόρεσα να τα συζητήσω όλα αυτά και έγραψα σε πολλούς από σας και προσβλέπω πάρα πολύ στις συζητήσεις και ερωτήσεις εδώ τις επόμενες εβδομάδες ίσως και πριν τα Χριστούγεννα. Ambassador, thank you for your uh, comment. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ευχές σας βέβαια και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε κάνει όλα αυτά τα σχόλια. Το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δίνω το λόγο στον κύριο Αλέν Καντέκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ για την υποδοχή στην Επιτροπή σας. Και θέλω να λάβω το λόγο ως πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας και σας αναφέρω την ομοφωνία της, ε, των μελών της Επιτροπής ε, Αλίας. Και έχω ήδη υποδεχτεί την ε, κυρία πρέσβη της των Φιλιππινών εδώ. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε στην στις Φιλιππίνες ότι μπορούν να θεωρηθούν ως τρίτη χώρα η οποία δεν συνεργάζεται ε, έναντι της ε, παράνομης και άναρχης αλίας. Με το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων για την, τις Φιλιππίνες. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα αλίας μπορούν να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμολογική επιβάλληση. Το GSP2 είναι μια εξαίρεση στους κανόνες του ΠΟΕ και επιτρέπει την είσοδο προϊόντων με δασμούς μηδενικούς. Εδώ πρόκειται και για προϊόντα της αλίας από τις Φιλιππίνες. Οι συντονιστές τη Επιτροπής Αλίας δεν δέχονται αυτήν την ε, εξουσιοδότηση πράξη για λόγους στους οποίους θα σας εξηγήσω. Η Κομισιόν έκουρσε τον κόδωνα του κινδύνου με την κίτρινη κάρτα που έδωσε στην, ε, στις Φιλιππίνες για την άναρχη και παράνομη αλία. Τόνισε την ανάγκη σεβασμού του ελέγχου και της νομοθεσίας για τον έλεγχο, γιατί δεν μπορεί κανείς να αποδείξει από τις Φιλιππίνες ότι τα προϊόντα αυτά που προέρχονται από τις Φιλιππίνες δεν είναι προϊόντα άναρχης και παράνομης αλίας. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές έναντι της παράνομης αλίας. Αν δεχτούμε όμως αυτή την πρόταση της Κομισιόν για κατεξουσιοδότηση πράξης, θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μια, έναν ανταγωνισμό από προϊόντα που δεν μπορεί να γίνει, να αποδειχθεί η προέλευσή του από νόμιμη αλία. Αυτό είναι αθέμητο ανταγωνισμό και το Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμα του 2011 ζήτησε να απαγορευτεί η πρόσβαση στην αγορά όλων των προϊόντων που προέρχονται από άναρχη και ε, παράνομη αλία και ζήτησε να σταματήσει η εμπορία προϊόντων που προέρχονται από τέτοια μορφή αλίας. Ούτω εχόντων των πραγματών, αν δεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα το σύστημα GSP για τις ε, Φιλιππίνες, για αύριο μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν είμαστε ενάντι, αλλά τώρα στις τωρινές συνθήκες θα γίνει δεκτό να μπει το, οι Φιλιππίνες στο σύστημα GSP πρέπει να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις ευθύνες του, γιατί οι Φιλιππίνες δεν τηρούν τους κανόνες για την παράνομη αλία ενώ θέλουμε να υπάρχει ένας τρόπος να είναι υπεύθυνα τα κράτη για την προέλευση των αλληλευτικών προϊόντων, αυτό θα επέτρεπε στις Φιλιππίνες να κάνουν το αντίθετο. Η συμπερίληψη λοιπόν των Φιλιππινών στο σύστημα GSP2 συν θα δημιουργούσε προβλήματα για τους αλληλείς τόνου. Αυτή τη στιγμή οι Φιλιππίνες είναι η κυριότερη ε, χώρα εισαγωγής για τα προϊόντα τόνου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν θα οδηγούσε στον παραλογισμό. Είπε η Κομισιόν ότι για λόγους μη διακρίσεως δεν είναι δυνατόν να εξαιρέσουμε τα προϊόντα λίας από το σύστημα GSP συν. Δεν υπάρχει κάποια λύση. Το είπε η Κομισιόν. Η Επιτροπή Αλίας όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελε να υπάρχει το... να υπάρχουν τα πορίσματα της δράσης της Κομισιόν, του σχεδίου δράσης της Κομισιόν για το σύστημα καταπολέμησης της παράνομης αλίας, προτού ξέρουμε ποια θα είναι η θέση μας για τις Φιλιππίνες και το GSP συν. Γι' αυτό ζητούμε από την Επιτροπή σας να πείτε όχι στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Δυστυχώ έχουμε και ένα πρόβλημα χρόνο διαγράμματος. Πρέπει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου να διατυπωθεί αυτή η αντίρρηση. Και στην Ολομέλεια πρέπει να γίνει αυτό μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Μα τα σχέδια το σχέδιο δράσης για την παράνομη αλία θα είναι γνωστό μάλλον στις αρχές του 2015. Θεωρεί η Κομισιόν ότι εμείς θα πρέπει να διαχωρίσουμε την εφαρμογή του κανονισμού έναντι της αλίας της παράνομης από την ε, προσχώρηση στο σύστημα GSP. Αυτό δεν γίνεται γιατί για ένα μεγάλο διάστημα θα μπορούν να μπαίνουν στην αγορά προϊόντα που πρόκειται από παράνομη αλεία. Έχουμε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, το καθήκον να εξασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσωτερική αγορά, πολιτική ανάπτυξη, πολιτική αλίας. Πρέπει να έχουμε κάποια συνέπεια με τον εαυτό μα. Δεν μπορούμε να λέμε κάτι και μετά να κάνουμε το αντίθετο. Δεν θέλουμε να πληττόμαστε από την ασυναρτησία σε αλληλευτική πολιτική και πολιτική εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο παρελθόν η αλληλευτική πολιτική ήταν ένας μπαλαντέρ της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να δεχτούμε αυτή την κατεξουσιώτηση πράξη, κατά την απόψή μου, είναι σαν να ψηφίζουμε με κλεισμένα τα μάτια υπέρ ενός υποψηφίου που δεν ξέρουμε το εκλογικό του πρόγραμμα. Θα ήταν μια τύφλη γκαβή απόφαση. Ω εκ τούτου θα ήταν καλύτερα και προ το συμφέρον τη ευρωπαϊκή Ένωσης να τροποποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για να λυθεί πρώτα το πρόβλημα της παράνομης αλίας και εφόσον λυθεί αυτό το πρόβλημα μπορούμε να εξετάσουμε την προσχώρηση των Φιλιππινών στο GSP συν. Σε αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή Αλίας θα υποστηρίσει απόλυτα και ένα ε, ψήφισμα το οποίο θα διατυπώνει αντίρρηση από το, την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτήν την θέση ομόφωνη της Επιτροπής Έλληνας. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη όπου έχουμε και ε, μέλη που καλούνται. Οπότε θα προχωρήσω ως εξής. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στις ε, πολιτικές ομάδες, στη Διεθνή ε, Επιτροπή Εμπορίου, μετά στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και έπειτα στους ευρωβουλευτές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής μας, αλλά έχουν προσκληθεί σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Ο κύριος Κασπάρη έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω μόνο να καταστήσω σαφές ότι τώρα δεν μιλάω εξ ονοματός μου προσωπικά, αλλά του κυρίου Φιέλνερ, που είναι ε, ο εισηγητής για το GSP, όπως ξέρετε. Και παραθέτω την γνώμη του. Ως εισηγητής για το βασικό κανονισμό περί GSP, ε, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί μου ε, την γνώμη μου μαζί σας τη γνώμη μου για το GSP. Καταρχήν, συμμερίζομαι τις ανησυχίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα της ε, βιομηχανίας αλληλείας. Ε, πρέπει αυτό πολύ σοβαρό να το λάβουμε υπόψη και γι' αυτό καλωσορίζω την έρευνα που έχει ξεκινήσει από την ε, αρμόδια γενική διεύθυνση ώστε να εξετάσει την μη αναφερόμενη και μη ρυθμιζόμενη αλληλεία. Είναι καθήκον της Επιτροπή αυτή να προσέξει και να ελέγξει κάθε νομικό θέμα που μας παρουσιάσει η Κομισιόν. Θα ήθελα να τονίσω την ε, νομιμότητα της ε, πράξης, καθώς και το ότι οι διάφορες υποψήφιες χώρες ε, που ετώνται αυτό το αίτημα, το καθεστώς θα πρέπει να, αν συμφωνούν με τα, αν τα κριτήρια, να το εκχωρήσει η Κομισιόν. Γιατί διαφορετικά δεν εφαρμόζεται ο βασικός κανονισμός σωστά. Δεν μπορεί δηλαδή μια απόφαση να βασίζεται μόνο σε, προσω... σε εκτιμήσεις, αλλά μόνο σε ρητή αναφορά στον κανονισμό διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων ήρθα σε επαφή με εκπροσώπου ε, των Φιλιππινών αλλά και εκπροσώπου ανθρωπιστικών οργανώσεων γιατί θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικά θέματα και να βρούμε άλλου τρόπου να αντισταθούμε στην κατεξουδότηση πράξη. Το θέμα είναι πω οι Φιλιππίνες τώρα δεν έχουν υπογράψει τις 27 ε, συμβάσει. Θα πρέπει να δούμε ωστόσο ότι ο κανονισμό λέει πω για να κερδίσει ειδικέ προτιμήσει η χώρα θα πρέπει να υπογράψει δεσμευτική ε, υποχρέωση για σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων, σεβασμό του περιβάλλοντος κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για αναπτυσσόμενες χώρες που δεν είναι τόσο τέλειος όσο εμείς, αλλά προσπαθούν να αναπτυχθούν όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Και γι' αυτό τους δίνουμε ένα, προ, ένα ε, κίνητρο για να εφαρμόσουν τις 27 συμβάσεις. Δηλαδή υπάρχει διαφορά μεταξύ της εισόδου στο GNP-SIN <coughs> γιατί και, και της ε, απλής γιατί μετά τη συνυπογραφή θα πρέπει να αποδείξουν οι χώρες ότι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές γιατί διαφορετικά μπορεί ε, να αποσυρθούν οι προτιμήσεις κάτι που συνέβη με τη Σρι Λάγκα πριν από λίγο καιρό. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα της ε, παράνομης ε, αλίας πολύ σοβαρά, γιατί εάν δεν είναι επιθυμητέ, ε, βιώσιμη η αλία, τότε μπορεί να υπάρξει, να ισχύσει ο μαύρος κώδικας, δηλαδή και να απαγορευτεί η αλία. Πρόκειται λοιπόν για έναν κανονισμό όπου πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Κομισιόν θα μπορεί να τον τηρήσει και εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να ζητήσουμε λογαριασμό από την Κομισιόν ε, και ελπίζω πως ε, η Φιλιππή, ότι δεν θα χρειαστεί να θεωρήσω υπεύθυνη την Κομισιόν ε, ότι δεν ανταποκρίθηκε στον κανονισμό. Και τώρα θα τα πω γερμανικά γιατί τώρα μιλώ εκ ονόματος της ομάδας μου ολόκληρης. Ποιο είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα ως προς τη χορήγηση του καθεστώτος GSP Plus στις Φιλιππίνες. Μπορούμε να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα της αλληλείας και δύο-τρεις εβδομάδες μετά να το αρνηθούμε. Μας λέει η Κομισιόν ότι από τη στιγμή που χορηγείται το καθεστώς αυτό μπορεί να αναθεωρήσει για τα ε, αλληλευτικά συγκεκριμένα. Η ομάδα μου ενδιαφέρεται πολύ να είναι πιο καλά οργανωμένα τα πράγματα από την πλευρά της των Φιλιππίνων για την αλληλεία και ενθαρρύνει την Κομισιόν να συνεργαστεί περισσότερο με τις αρχές των Φιλιππίνων για να υπάρξουν βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Έρχομαι τώρα στους σοσιαλιστάς. κυρία Μόσκα. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν που είναι σήμερα εδώ και που μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους ε, καταρχήν το γεγονός ότι αυτή η εκχώρηση του προτιμησιακού συστήματος για τις Φιλιππίνες θα είναι η πρώτη για αυτό το νέο θητεία του Νέου Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίο μας επιβαρύνει με μεγαλύτερη ευθύνη διότι δεδομένων των επίμαχων σημείων για τα οποία συζητάμε, μας επιβάλλεται μια λεπτότητα, μια ευαισθησία που θα συνεχιστεί και στην υπόλοιπη εντολή. Εγώ λοιπόν ε, συμμερίζομαι αυτή την ανησυχία καταρχήν γιατί πρέπει να δείξουμε την συνέπειά μας αλλά και την, το κατά πόσο είμαστε ε, αξιόπιστοι σε σχέση με ρυθμιστικές δοκιμές που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε αυτό το προτιμησιακό καθεστώς τη στιγμή που καλύπτονται όλες οι απαραίτητες ε, προϋποθέσεις. Ωστόσο, υποστηρίζω επίσης τη θέση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί ως βραβείο. Αντίθετα, είναι μια ευθύνη. Ε, στις οποίες, γιατί στις χώρες στις οποίες χωρούμε το προτιμησιακό καθεστώς θα πρέπει να τον αναλάβουν αυτή την ευθύνη γιατί ξεκινά μια πορεία έτσι. Σε αυτή τη νέα φάση της ε, υπερορικής πολιτικής που ξεκινάμε πιστεύω πως είναι σημαντικό να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το πέρασμα έτσι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν αυτά τα το καθεστώτα χωρίς ταυτόχρονα να γίνεται πολύ έντονη παρακολούθηση. Από μια πλευρά λοιπόν υπάρχει η ευθύνη από πλευρά των χωρών στις οποίες ε, χωρείται αυτό το σύστημα, από την άλλη όμως υπάρχει η ευθύνη η δική μας και της Κομισιόν, έτσι ώστε να γίνεται παρακολούθηση εξ αρχής πολύ στενή, κυρίως για τα πιο λεπτά ζητήματα και ε, με βάση αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα ακόμα και στην περίπτωση που, για την οποία μιλάμε και πρέπει λοιπόν να στηριχθεί να στηριχθούν όλες οι δράσεις ε, παρακολούθησης που θα στηρίξει η Κομισιόν στη νέα φάση ε, δεδομένης της ποσότητας του όγκου των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια τέτοια ε, ανάλυση, να δούμε ποιοι είναι οι πόροι μας, ώστε να γίνεται ε, πιο στενή παρακολούθηση. Πολύ περισσότερα από όσα έχουν γίνει στο παρελθόν. Για να φτάσουμε τώρα στο θέμα του ερωτήματος για την αλληλεία, που είναι ακριβώς το πιο λεπτό ε, ζήτημα εμπορικά, θεωρώ ότι σε στο πνεύμα των όσων είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, να πρέπει να εγγυηθούμε ναι τη συνέπεια, αλλά να μπορούμε να προχωρήσουμε σε παράλληλους δρόμους και άρα να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση στην αποδοχή της πρότασης να επιτραπεί το προτιμησιακό αυτό καθεστώς, αλλά να μην υπάρχει καμία, κανένας περιορισμός σε περίπτωση που χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πιο αυστηρή εκτίμηση, φτάνοντας και σε μια πιο έντονη ε, διαδικασία, πούμε, να δώσουμε κόκκινη κάρτα, εάν ε, δεν ε, τηρηθούν απόλυτα ή τα προποτήμενα από πλευράς των Φιλιππινών. Πιστεύω λοιπόν πως το ίδιο το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να σεβαστεί την συνέπεια και θα πρέπει μάλλον να σεβαστεί τη συνέπεια και την αξιοπιστία και να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. For the conservatives, uh, our colleague McClarkin. Η κυρία Μακλάρκιν από τους συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον πρέσβη που ήρθε σήμερα εδώ και μας ε, τόνισε πόσο, σημαντική είναι, ε, πόσο σημαντικό είναι το καθεστώς ε, του πρωτομενησιακού για τον λαό των Φιλιππινών. Σημαίνει ότι εμείς, εμείς έχουμε στηρίξει τις Φιλιππίνες και για το προτιμησιακό καθεστώς και για το GSP Plus που ε, θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Η αλληλευτική βιομηχανία δεν είναι τμήμα των κριτηρίων και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ενθαρρύνω τον πρέσβη να διαβιβάσει αυτό το μήνυμα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το καθεστώς και για μας και να πω και στην Κομισιόν ότι η στεναρή παρακολούθηση αυτού του καθεστώτος είναι απαραίτητη και ότι πρέπει να τρίσουμε τους κανόνες, να έχουμε αυστηρούς κανόνες, να τα έχουμε, τους έχουμε, αν πληρώνται τα κριτήρια να προχωρήσουμε. Πάντως, όταν έχουμε ας πούμε κίτρινη κάρτα θα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε την θέση μας. Θέλω αυτά τα μηνύματα να περάσω στη Ευρωκομισιόν και στον Πρέσβη και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του GSP. Συν. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Σάκε για την άλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, κυρία Πρέσβη για, τον, κόσμο των Φιλιππινών πολύ περιμένουν αυτό το καθεστώς. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της χώρας επί τη βάση ο, κανόνων και όχι μόνο στην οικονομία αλλά και όσον αφορά την προοπτική της χώρας. Το νέο σύστημα GSP είναι πιο αυστηρό αλλά περιλαμβάνει και διατάξεις για την παρακολούθηση. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να επαληθεύει την ανταπόκριση στα κριτήρια και την συνυπογραφή των 27 διεθνών συμβάσεων για την παιδική εργασία, το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, ελεύθερης έκφρασης και είναι θέματα που μας είναι μας πολύ ε, προσφυλή. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση. Όμως θα πρέπει ε, να τηρήσουμε τους κανόνες γιατί ο GSP. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Τα ακούσαμε και από την κυρία Πρέσβη. Να είμαστε βέβαιοι πώς θα, θα εξετάζει πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις. Και ότι όλα αυτά θα γίνονται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ. Και το Άγιο είναι πολύ σημαντικό και πολλοί το ανέφεραν. Παράνομη και μη ρυθμιζόμενη ελεία αλλά Πιστεύουμε πως τα δύο αυτά θέματα, δηλαδή το IUU και η παρακολούθηση του αλλά και την παρακολούθηση των, ε, του καθεστώτος γενικευμένων προτεμήσεων είναι χωριστά θέματα. Η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσει ανεξάρτητα από το αν χορηγηθεί το καθεστώς ε, GSP, να προχωρήσει απέναντι στις Φιλιππίνες αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, για παράδειγμα απαγόρευση των εισαγωγών. Ωστόσο είναι δύο διαφορετικά ζητήματα και εδώ και δεν είμαστε αντίθετοι αυτή τη στιγμή σε κατεξιοδότηση πράξη. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Όχι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την κατάσταση για τις Φιλιππίνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί έχει πολύ κακή φήμη η χώρα αυτή. Είναι μια από τις πέντε χώρες όπου η Διεθνής Αμνηστία στόχευσε την πρόσφατη της εκστατεία κατά των μαρτυρίων, των βασανιστήριων, γιατί αυτά ανθούν στις Φιλιππίνες. Δεν αρκεί να συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να μιλήσουμε για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για προτιμησιακά τέλη. Και αυτό σημαίνει διαρκή παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Η Κομισιόν συμφωνεί μαζί μου και αν ναι, πώς θα καταστούν τα ανθρωπίνα δικαιώματα κατευθυντήρια αρχή Τώρα, από την άλλη πλευρά δεν πρόκειται όλα να γίνουν ρόδινα μόλις γίνει αυτή η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Απλά ανησυχούμε για τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου για τους αλληλείς καταρχήν αλλά και για το περιβάλλον. Κάποιοι συνάδελφοι γρήγορα, γρήγορα αρχίζουν και δημαλώνουν τις άλλες χώρες όταν προσπαθούν να προστατεύσουν τις αγορές τους, αλλά σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ελευτική Βιομηχανία θα πέσει και θα πλακώσει την Φιλιππινέζικη Ελευτική Βιομηχανία. Ποιο ήταν ο αντίκτυπος αυτή τη συμφωνία για την οικονομία και το περιβάλλον των Φιλιππινών. Και επίσης οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι που πιέζουν για τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις ε, δεν πιέζουν αν ναι, ποια είναι τα αιτήματά τους. Ευχαριστώ. Ε, going to the... Ευχαριστώ. Πηγαίνω στους πράσινους. Ο κύριος Ζαντό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντυπωσιάζομαι από το ύφο ορισμένων παρεμβάσεων που είναι σαν να λένε ότι το θέμα της παράνομης αλληλείας, της μη υποκείμενους σε κανόνες, δεν είναι σημαντικό ή σοβαρό ή μια τυπική υποχρέωση για να αποκτήσει κανείς το καθεστώς GSP συν, οπότε ας συνεχίσουμε για τα εμπορικά θέματα και το θέμα αυτό της αλίας να το αντιμετωπίσουμε σε άλλο χώρο. Όταν το 1 έκτο των εισαγωγών στην Ευρώπη από τις Φιλιππίνες είναι προϊόντα αλίας για τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία για πρακτικές οι οποίες είναι τελείως παράνομες και δεν υπόκεινται σε κανόνες, εγώ δεν καταλαβαίνω την συνεκτικότητα των λόγων ορισμένων συναδέλφων. Καταλαβαίνω ότι οι Φιλιππίνες έχουν δεσμευτεί να υπογράψουν μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις και αυτό είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την ε, απονομή του καθεστώτος GSPC αλλά δεν λέτε τίποτα για την ποιότητα των εισαγωγών από τις Φιλιππίνες και ιδίως από τη στιγμή που σήμερα οι Φιλιππίνες είναι μέσα στις χώρες οι οποίες ακολουθούν την ε, παράνομη και άναρχη αλληλεία. Δεν νομίζω ότι σήμερα έχει νόημα να τους δώσουμε το καθεστώς αυτό του GSPC. Για μας ως πρασίνους το θέμα δεν είναι να εμποδίσουμε τις Φιλιππίνες να έχουν αυτό το καθεστώς, κάθε άλλο αλλά όσο παραμένει το πρόβλημα αυτό της παράνομης και δεν έχει επιληθεί θα είναι τελείως χωρίς λογική να δώσουμε αυτό το καθεστώς στις Φιλιππίνες. Ευχαριστώ πολύ για την EFTD. Ναι παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μετά από αυτά που είπε ο κ. Ζαντό και εγώ ίδια θεωρώ ότι είναι παρά, απαράδεκτο να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Χωρίς να έχουμε μια απόλυτη εγγύηση για την θέση ε, για την, ε, και τις, τις επιπτώσεις στην αλληλεία των Φιλιππινών. Δεν έχω άλλο κάτι να πω. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε συναδέλφους που θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι πολύ σύντομοι στις ε, παρεμβάσεις τους. Καταρχήν ο Γέρος Λαβαλέσα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα κάποιους ε, που προσπαθούν να χωρίσουν ε, την αλληλεία από το πακέτο. Δεν πρέπει ποτέ να το εξετάσουμε ως χωριστό θέμα. Και αν ναι, τότε είναι αποτυχία αυτό. Να σας θυμίσω το άρθρο 9β του κανονισμού GSP καθιστά ερετούς, ερετά τα, τα ωφέλη το GSP+. Plus. Μόνο τα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα δικαιολογήσει, αιτιολογήσει την αναστολή μιας τέτοιας ε, συμφωνίας και νομίζω πως ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ε, το θέμα αυτό ως ένα πακέτο, μια δέσμη και να μην ξεχωρίσουμε την ελευτική βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω την πρέσβη της Φιλιππίνες και να υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή μας συνεργάζεται με τη νέα Επιτροπή Juncker και ελπίζω ότι αυτό που είδαμε σήμερα δεν είναι προηγούμενο για τις μεταγενέστερες συνεδριάσεις μας. Ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με την ε, Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Για το ζήτημα τώρα το οποίο μας απασχολεί. Θέλω να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Μιλάμε για ένα θέμα όπου δεν νομίζω ότι κανείς έχει κάποια αντίρρηση το να υπάρχει ένα σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για τις Φιλιππίνες. Νομίζω ότι έχουν γίνει σεβαστές όλες οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι Φιλιππίνες στο σύστημα αυτό και υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα. Από τις 13 χώρες οι οποίες είναι αντικείμενο αυτού του συστήματος είναι ορισμένες οι οποίες έχουν δεχτεί μια κίτρινη κάρτα παραβιάζοντας τη διεθνή νομοθεσία. Αυτά τα οποία θεωρεί δηλαδή παράνομα η Κομισιόν για την αδήλωτη και παράνομη αλία. Όχι, εδώ λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μια τελείως εξαιρετική κατάσταση και η οποία έχει τεράστια σημασία για την αλληλευτική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες εξαρτώνται από την αλληλεία. Έχουν λοιπόν παραταθεί οι προθεσμίες, αλλά αυτή τη στιγμή, αν προχωρήσουν όλα όπως ε, προβλέπονται, θα γίνει ψηφοφορία το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα πρέπει να περατωθεί το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, σαν αποτέλεσμα της κίτρινης κάρτας που έχει δείξει στην Κομισιόν, η, στις Φιλιππίνες η Κομισιόν. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τον Ιανουάριο για να ξέρουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως αναρωτιέμαι αν μπορούμε να δώσουμε προτιμήσεις στο χρονοδιάγραμμα ή αν θα θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε τους στόχους που όλοι ενστερνιζόμαστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προύστη ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε συνάδελφοι, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας Αλεν Καντέκ, υπάρχει ένα θέμα χρονοδιαγράμματος εδώ και όλα τα νομικά επιχειρήματα δεν μπορούν να απαντήσουν στο θέμα της πολιτικής αξιοπιστίας. Δεν μπορώ ως Ευρωβουλευτής να εγκρίνω την εισαγωγή αλλιευμάτων που προέρχονται από παράνομη αλληλεία. Και αυτό το θέμα της αξιοπιστίας δεν λύνεται με κανένα νομικό τρόπο. Γι' αυτό προτείνω να μπλοκάρουμε την ένταξη των Φιλιππινών στο GSP συν όσο δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εξάλλου και άλλοι είπαν ότι οι Φιλιππίνες ε, φυσικά μπορούν να ξαναζητήσουν ένταξη στο, τα μέσα του επόμενου έτους όταν θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένας κατεπήγον χαρακτήρας για να εγκριθεί αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη. Ενώ υπάρχει ένα επιχείρημα για την απόρριψη ότι δεν θα υπάρξει εγγύηση ότι αυτά τα αλλιεύματα που θα εισαχθούν θα είναι νόμιμα. Η Κομισιόν μας είπε μηχανικά αυτά που μας απάντησε και γραπτός. Το θέμα της παράνομης αλληλείας δεν εξαρτάται από τις υποψηφιότητες στο σύστημα GSP-SYN. Παρόλα αυτά το gsp μπορεί να είναι ένα εργαλείο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα των 27 συμβάσεων που συνδέονται με το GSP συν. Η Κομισιόν θεωρεί ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι από το προηγούμενες επικρίσεις του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του, του 12 που καταδίκαζε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες. Η Διεθνής Αμνηστία προετοιμάζει εξάλλου ένα ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες το Δεκέμβριο. Αν η έκθεση αυτή είναι πολύ επικριτική που είναι το πιθανότερο σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε πώς θα αντιδράσει, πώς θα δικαιολογήσει η Κομισιόν τον επόμενο μήνα στις, μπροστά στις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις την έγκριση αυτών των 27 συμβάσεων από τις Φιλιππίνες. Ας μιλήσουμε και για την εξισορρόπηση της κατάστασης στην Νοτιοανατολική Ασία. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη, ιδιαίτερα για τον Ανανά αν μια γειτονική χώρα εξάγει με δασμό 0% το ίδιο προϊόν που εκείνες εξάγουν με 18 και 14% δασμούς. Αυτή η ανισορροπία δεν θα θέσει προβλήματα για τις γειτονικέ χώρες των Φιλιππίνων σε ορισμένους τομείς. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω εδώ μια αντίφαση. Μία από τις 27 συμβάσεις αφορά την ελάχιστη ηλικία των εργαζομένων και έχει εγκριθεί από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο το 2013 σημείωσε ότι περίπου 550.000 ανεξάρτητων εργαζομένων στις Φιλιππίνες είχαν ηλικία 5 με 17 ετών και αυτό σε κατάφορη παραβίαση της σύμβασης. Πώς μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να θεωρεί ότι οι συμβάσεις αυτές εφαρμόζονται όλες σωστά ενώ η κύρια οργάνωση που αφορά θέματα εργασίας βρίσκει παραβιάσεις για τις Φιλιππίνες αυτό το θέμα θέτει πολλά και λεπτά ερωτήματα. Επομένως δύο, διήν θάτερον. Τα δύο ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα. Μπορούμε να εγκρίνουμε την εισαγωγή αλλιευμάτων χωρίς να είναι εγγυημένη η προέλευσή τους, αν είναι νόμιμη ή παράνομη. Και δεύτερον, θέλουμε το GSP να γίνει ένα εργαλείο με προώθηση, με παρότρινση, αλλά Ποιος θα παροτρύνει αυτή η ένταξη. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να εγκρίνω ούτε μπροστά στα μάτια των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ούτε μπροστά στα μάτια των οργανώσεων των αλλιών, γιατί πρέπει οι Φιλιππίνες αυτή τη στιγμή να ενταχθούν στο GSP+. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Μπλάνκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να ακούσω διαφορετικές απόψεις οι οποίες αναφέρονται στην εφαρμογή μιας πράξης κατά που θέτουν πάρα πολλά ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, είμαι μέλος της Επιτροπής Αλίας και εγώ χρειάστηκε να φύγω από την Επιτροπή Αλίας για να είμαι εδώ παρόν. Μιλάμε πράγματι για ένα ζήτημα το οποίο έχει μια σημαντική σημασία για κάποιες από τις περιοχές μας και ιδίως για τη Γαλλικία που είναι μία από τις πιο σημαντικές αλληλευτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ υπάρχει η πρόταση να εγκρίνουμε μία απόφαση χωρίς να λάβουμε υπόψη τις ε, συνέπειες της ε, έγκρισης αυτής για την ε, βιομηχανία κονσέρβα τόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο κατά την άποψή μου δεν μπορεί να τύχει απόφαση χωρίς να λάβουμε υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της απόφασης. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά βέβαια, όπως ξέρετε, ότι καταρχήν η Κομισιόν θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση αν δεν έχουμε το Δεκέμβριο μια έκθεση η οποία καταδεικνύει όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και των αρχών της ευκυβερνησίας που είναι απαραίτητη να ισχύουν για να πάρει μια χώρα το καθεστώς του GSP συν. Επίσης θα ήταν πολύ αρνητικό τη στιγμή που υπάρχει μια κίτρινη κάρτα για τις Φιλιππίνες ήδη σε σχέση με τις εκθέσεις οι οποίες διατυπώνονται και οι οποίες αναφέρουν ότι οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα που δεν έχει συνεργαστεί μαζί μας σε σχέση με την παράνομη αλία. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή προτείνουμε μια λήψη απόφασης η οποία είναι δεδιασμένη, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις και με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με ζημίες που μπορούν να προκύψουν για περιοχές όπως η Γαλλικία και που μπορεί να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα εάν εφαρμοστεί αυτή η άνηση μορφή ανταγωνισμού με τις Φιλιππίνες. Κανείς δεν έχει πρόβλημα με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε δεδομένο, αλλά θα πρέπει να καθορίζονται οι συνθήκες ανταγωνισμού και αν δεν υπάρξει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων και αν επιπλέον υπάρχουν στοιχεία ε, υποψίας σε σχέση με το πώς γίνεται η αλία και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνεται με τρόπο ο οποίος είναι παράνομος και δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε κάνουμε πραγματικά ένα μεγάλο λάθος και δεν βοηθάμε τις δικές μας επιχειρήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύω πρέπει να το δεχτούμε όχι μονάχα για την τον αλληλευτικό κλάδο, αλλά σε ό,τι αφορά και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Χαίρομαι λοιπόν το ότι ήδη σε αυτή την Επιτροπή υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ανησυχίες για αυτό το θέμα. Εμείς νομίζαμε ότι αφορούσε μονάχα τους αλληλείς, αλλά βλέπω ότι ευτυχώ ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αντίθετοι και χαίρομαι για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μας έχει μια ζωντάνια. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, uh, Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μιλάν Μον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την ε, πρέσβη των Φιλιππινών που είναι παρούσα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή Αλία και όπω είπε ο πρόεδρό μα, <clears throat> ο κύριο Καντέκ, επειδή έλαβε το λόγο, δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μπει στο GSP οι Φιλιππίνες, ενώ συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε τη λεγόμενη κίτρινη κάρτα στις Φιλιππίνες και τους απειλεί με απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων αλίας αν δεν σεβαστούν τους κανόνες για την άναρχη και παράνομη ε, αλία. Είναι κάπως αντιφατικά αυτά. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είχαν για τις Φιλιππίνες. Θα έπρεπε να μου πει η Κομισιόν αν υπήρξε κάποια πρόοδος στις Φιλιππίνες στον αγώνα εναντίον της παράνομης, της αδήλωτης και ε, ακανόνιστης αλίας. Είχα ρωτήσει την Κομισιόν αν υπάρχουν ε, πρόοδοι, αλλά δεν έχω πάρει απόφαση. Ανεξάρτητα από το GSP συν για τις Φιλιππίνες, θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να λάβει κάποια μέτρα αν δεν υπάρχει πρόοδος για την πάταξη αυτής της παράνομης αλίας της Φιλιππίνες και κρατήσει κάποιο παραλληλισμό για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά στη δική μου περιοχή, την Γαλλική, από την οποία προέρχεται και ο κύριος Μπλάνκο, όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή κονσερβοποιημένου τόνου που μπορεί να θυγεί από την άρση των δασμών για την, ε, τις Φιλιππίνες και πάρα πολλοί παραγωγοί βλέπουν με εμβρόντιτο τρόπο πως μια χώρα που δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μια ελεύθερη δασμόν εξαγωγή αλληλευτικών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει και να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Μια αίτηση ακόμα για να λάβει κάποιος το λόγο δεν ξέρω εκτό από την κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ αν θέλει να λάβει κάποιο το λόγο. Κλείνω τον κατάλογο των αγωγητών και δίνω το λόγο στην Βίβιαν Ρέντινγκ. Ναι, Πρόεδρε. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι από τη μία έχουμε το σύστημα γενικημένων προτιμήσεων ΣΥΝ με τα κριτήρια του και τα κίνητρα που δίνει με στόχο να ξεπεράσουμε τη στεγνή οικονομική διαχείριση γιατί οι Φιλιππίνες θέλουν να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό και για τις Φιλιππίνες και για την Ευρώπη ολόκληρη. Πρέπει βέβαια να υπάρχει μια συνοχή στην εφαρμογή όλων αυτών των σχεδίων και πολύ σοβαρή εποπτεία από την Κομισιόν. Άκουσα επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο συνάδελφος Βαλέντσα για τους όρους που εγγράφονται στο σύστημα. Απ' την άλλη, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που το εξήγησε πολύ καλά ο συνάδελφός μας από την Επιτροπή Αλίας όπου έχει δοθεί κίτρινη κάρτα. Έχει γίνει μια έρευνα με κατηγορία παράνομη αλία. Μπορούμε λοιπόν εμείς τώρα να έρθουμε σε αντίφαση με τους εαυτούς μας, δηλαδή να δώσουμε την άδεια για μια ένταξη η οποία σημαίνει ότι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα, μπει η θα μπουν οι Φιλιππίνες στο πρόγραμμα και ταυτόχρονα να συζητιέται η έρευνα παράλληλα. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας και ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια ασυνέπεια στην πολιτική μας δράση. Ιδίως διότι είναι και πολύ κοντά όλα αυτά χρονικά. Κοντά. Ευχαριστούμε. Και για να συνοψίσουμε τώρα θα ήθελα να στραφούμε προς την πρέσβυρα των Φιλιππίνων εάν νομίζει ότι χρειάζονται ορισμένες απαντήσεις. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι και μετά θα μιλήσει πάλι η Κομισιόν. Ορίστε κυρία πρέσβυρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως χώρα που όπως και στις δικές σας εφαρμόζει το κράτος δικαίου, θα σας έλεγα να εφαρμοστούν οι κανόνες πρώτα-πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, δύο τρόποι υπάρχουν να το λύσουμε αυτό. Ο ένας είναι ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Μόνς. Να ζητήσουμε από την Κομισιόν, να ρωτήσουμε την Κομισιόν τι γίνεται στο διάλογο μας για αυτή τη λεγόμενη κίτρινη κάρτα δεν είναι κόκκινη στο κάτω-κάτω, κίτρινη είναι. Σημαίνει ότι μπορεί η χώρα να μην συμμορφώθηκε σε όλα πλήρω. Υπάρχει μια εξάμεινη διαδικασία που προβλέπετε και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω περαιτέρω πληροφορίες, αλλά υπάρχουν 12 σημεία που δέχτηκαν οι Φιλιππίνες που συμφώνησαν με την Κομισιόν και από αυτά τα 12 έχουν όλα σχεδόν πληρωθεί. Το μόνο που επικρέμαται ακόμα είναι δύο. Ένα, μία τροπολογία του αλλιευτικού κώδικα των Φιλιππίνων για την αύξηση των προστήμων για την παράνομη αλληλεία στην ανοιχτή θάλασσα. Δυστυχώς το Κογκρέσο των Φιλιππίνων ε, έχει διακοπές αυτή τη στιγμή αλλά θα ξαναγυρίσει στις 17 του μηνός και τον επόμενο μήνα θα υπάρχει ο νόμος δεύτερον Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα για την εποπτεία, για την αξιολόγηση, για τα VMS. Πρόσθετο προσωπικό 1.700 ατόμων για την επιτήρηση ακριβώς και τα λοιπά. Υπάρχουν όλα αυτά και σας συστήνω να τα εξετάσετε και τότε θα φανεί η λύση αμέσως λύγει το πρόβλημα, θα αφαιρεθεί η κίτρινη κάρτα μέχρι το τέλος του μήνα. Και τότε μπορείτε να ψηφίσετε για την ένταξή μας στο GSP+. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πρέσβυρα και τώρα η Κομισιόν και θα ήθελα να μας σχολιάσει σύντομα και το θέμα της κένειας της Κενίας μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να διαλύσω τους φόβους ότι έχουμε διασπασμένη, προδιχασμένη προσωπικότητα στην Κομισιόν. Εμείς δουλεύουμε με απόλυτη συνέπεια και συνοχή μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Καταρχάς το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως ο κανονισμός του GSP μας επιβάλλει συγκεκριμένες διορίες. Πρέπει μέσα σε έξι μήνες να αποφασίσουμε. Και σύμφωνα με τη διαδικασία λοιπόν αυτή πρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μετά σε άλλους τέσσερις μήνες να έχουν αποφανθεί. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Η αναβολή δηλαδή και η καθυστέρηση δεν γίνεται με βάση το κανονισμό. Θα ήταν παράνομο. Για μας λοιπόν το θέμα ότι τα δύο εργαλεία λίγο πολύ θα φτάσουν το Δεκέμβριο στο τέρμα τους, σωστό μου φαίνεται. Και καλό, θετικό. Θα απαρθεί η απόφαση για το GSP+, αλλά για την παράνομη αλληλεία, την οποία λέμε με άλλα λόγια στη γλώσσα μας IUU, δεν νομίζω ότι μπορεί σίγουρα να λυθεί σε ένα μήνα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το GSP είναι εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης ενώ η παράνομη αλληλεία κάτι συγκεκριμένο για την αλληλεία. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία και άλλα που εργάζονται παράλληλα. Παράδειγμα, οι διαδικασίες anti-dumping. Το GSP Plus δεν προσφέρει καμία προστασία ως προς όλα, σε σύγκριση με όλα τα άλλα εργαλεία για παράνομο εργαλείο. Έχουμε διαδικασίες anti-dumping από χώρες που ωφελούνται με το, από το BGSP Plus για τις Φιλιππίνες συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο ε, έγινε η πρώτη καταγγελία και δεν προβλέπεται καθυστέρηση της απόφασης για το GSP Plus εάν υπάρξει καταγγελία για κάτι σχετικά ε, αρκετά άσχετο. Είναι παράλληλα αυτά τα δύο. Αν ας πούμε υπάρχει περίπτωση anti-dumping ή dumping για την αλληλεία, τότε μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα σε σχέση με το αντι dumping ανεξαρτήτως από το καθεστώς GSP Plus ή όχι. Αντίθετα, νομίζουμε ότι η ανεξαρτησία των δύο εργαλείων είναι μια εγγύηση. Η παράνομη αλληλεία το ίδιο. Σας Βεβαιώνω λοιπόν ότι για το IUU, για την παράνομη αλληλεία, εάν τελικά χορηγηθεί κόκκινη κάρτα που δεν ισχύει σήμερα, τότε θα ληφθούν μέτρα. Το GSP Plus δεν θα προστατέψει τις Φιλιππίνες από αυτή τη διαδικασία. Έπειτα, κάποιος είπε ότι πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση. Είχα πει και προηγουμένως ότι πρέπει να δείχνουμε ισοτιμία και ισοψυχία Υπάρχει κι άλλος ωφελούμενος από το GSP Plus με την ίδια κατάσταση, με κίτρινη κάρτα. Και αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει το καθεστώς GSP Plus. Χαίρομαι γιατί η χώρα εκείνη είχε ακολουθήσει όσα του συνέστησε η Γενική Διεύθυνση Θαλασσιών Υποθέσεων και τώρα πήρε πράσινη κάρτα. Το ένα εργαλείο λοιπόν δεν εμποδίζει το άλλο. Τώρα για την ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα πράγματι είναι θέμα που λόγω του τρόπου που εγκρίθηκε ο κανονισμός δεν προβλέπει να κάνουμε ανάλυση για τη σχετική ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων προϊόντων. Και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Παρ' όλα αυτά, ο κανονισμός έχει μερικές ρήτρες που μας διασφαλίζουν στις περιπτώσεις αυξανωμένων εισαγωγών και τιμών κτλ. Υπάρχουν ρήτρες ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν εάν υποβληθεί δε δικαιολογημένη προσφυγή. Οι ειδικέ ασφαλιστικές ρήτρες λοιπόν για τη γεωργία και την αλληλεία είναι πιο αυστηρές από τις κανονικές εφόσον υποβληθεί δε δικαιολογημένη προσφυγή. Υπάρχει λοιπόν εδώ, έχουμε εργαλεία για δίκαιο εμπόριο για... και γι' αυτό οι ρήτρε ασφαλείας μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και αν δεν έχει διαπιστωθεί παράνομη πρακτική. Αλλά απλώς απρόβλεπτη αύξηση τιμών ή όγκων. Αν μπορεί αυτό να αποδειχθεί λοιπόν ότι δηλαδή δημιουργεί αυτό δυσκολία στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Τέλος για τις 27 συμβάσεις. Εδώ δεν επιβραβεύουμε χώρες που εφαρμόζουν τις συμβάσεις κατά 100% και χώρες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έχουν εφαρμόσει αυτές τις συμβάσεις και πολλές χώρες της Ένωσης και φυσικά οι αναπτυσσόμενες χώρες αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουν πολύ πιο δύσκολα. Σκοπός του εργαλείου λοιπόν είναι τα κίνητρα για να αρχίσουν να τα λύνουν αυτά τα προβλήματα και το GSP Plus έχει τις, εγγυήσεις, τις εποπτικές εγγυήσεις που το επιτρέπουν. Αυτά για το GSP Plus. Τώρα όμως θα ήθελα να μιλήσω για ε, μια διαφορετική ήπειρο για να αναφερθώ δηλαδή σε μια άλλη κατεξουσιοδότηση περίπτωση εκείνη που σχετίζεται με το GSP Plus και είναι εκείνη της Κενίας. Θα είδατε σε αυτή την Επιτροπή το Σεπτέμβριο ότι εγκρίθηκε μια κατεξοδιόμενη πράξη που έθεσε διάφορες ε, αφρικανικές χώρες ε, υπό το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων διότι θα έφευγαν από εκείνο το ΜΑΡ που ήταν μια άλλη ρύθμιση προτιμησιακής ε, ε, προτιμησιακού καθεστώτος. Όλε αυτέ οι χώρες εκτό από την Κένια προχώρησαν σε αυτά τα βήματα που έπρεπε για να επανεσωματωθούν στο ΜΑΡ. Η Κένια ήταν η μόνη από, που, μέχρι την πρώτη δεκάτου δεν το είχε πράξει γιατί αυτή ήταν η προθεσμία για το ΜΑΡ. Να σας πω λοιπόν τα καλά νέα ότι τώρα η Κένια μαζί με άλλες χώρες στην Αφρική ε, συνυπέγραψαν ε, ε, το EPA της Ανατολικής Αφρικής την Συμφωνία εταιρική Σχέσης και έτσι μπορεί να επανέλθει στο ΜΑΡ και αυτό θα σας ανακοινωθεί μόλις θα γίνει και επισήμως. Αυτό σημαίνει βέβαια πως όλες αυτές οι χώρες που υπόκειται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων επειδή όλες την χάνουν ε, μεταχείρισης ΜΑΡ θα απέρθουν από το σύστημα GSP όταν θα γίνει αναθεώρηση των δικαιούχων του χρόνου. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό το θέμα θα διοργανωθεί σε επόμενη ευκαιρία για την Κένια. Για την Κένια, όχι, αλλά, συγγνώμη, αλλά έχουμε αργήσει πάρα πολύ στην ημερήσια μας διάταξη και δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για την Κένια, αλλά θα μπει στην ημερήσια διάταξή μας και η Κένια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 Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Πριν έρθουμε στο σημείο 15, μια σύνομη παρατήρηση για το σημείο 9 της ημερησίας διάταξης, που είναι οι δασμολογικές ε, διατάξεις για το Εκουαδόρ. 6 Νοεμβρίου στις 18.00 το απόγευμα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες για το θέμα αυτό. αυτό. Έχουμε άλλα τρία σημεία τώρα στην μέση διάταξη και θέλω να σας παρακαλέσω για το τελευταίο σημείο που είναι το ζήτημα της συμφωνίας με την Σιγκαπούρη να έχουμε αρκετό χρόνο και θα πρέπει να διαλευκανθεί το θέμα του αν είναι μεικτή συμφωνία ή όχι αυτή με την ε, Σιγκαπούρη. Σημείο 15 λοιπόν. Συμφωνία σύνδεσης με τη Γεωργία. Ο Όλι Ρεν είναι ο εισηγητής μας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να θυμάστε ότι παρουσίασα τα βασικά στοιχεία για αυτό το ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα επανέλθω για την ουσία της συμφωνίας αυτής καθεαυτής. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης <clears throat> που αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί φαίνεται να ακολουθούν την γνωμοδότησή μας για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης της ε, Μολδαβίας στην προηγούμενη μας συνεδρίαση. Υπήρξαν τώρα πολλές τροπολογίες, οι οποίες γενικά βελτιώνουν το κείμενο, δίνουν μεγαλύτερη ειδικότητα στα ζητήματα αυτά. Βέβαια είναι ίσως κάπως πιο τεχνικές στη μορφή τους, και κάποιες από αυτές έχουν το χαρακτήρα συμβαστικών τροπολογιών και γι' αυτό θα να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους. Για τις τροπολογίες αυτές τώρα. Τόσο οι τροπολογίες Κάσπερι όσο και Λαντσμπέργκης υπογραμμίζουν τη σημασία του να γίνει κύρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ταχαίως και χωρίς περιττή καθυστέρηση ώστε να εφαρμοστούν οι οικονομικέ και εμπορικέ ρήτρε. Ο κύριος Φλαντσπέργης έχει, έχει <clears throat> υποβάλει και τροπολογίε για την ανάγκη να υπάρξει μεταλαμπάδευση τεχνολογία, οικονομικέ μεταρρυθμίσει και προσέγγιση τη νομοθεσία. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε γιατί πάντα δεν έχουμε απουσία δυσκολιών. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να αναπτύξει η γεωργία μια οικονομία της αγοράς. Για τις τροπολογίες του κυρίου Ζαχραουντόου, η τροπολογία 2 αναφέρεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η τροπολογία 4 υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της συμφωνίας ελευθέρω εμπορίου για τις μικρομεσαίες που θα οδηγήσουν σε ένα πιο προβλέψιμο ε, περιβάλλον για επενδύσεις. Υπάρχει και μια τεχνική τροπολογία του κυρίου Ζαχραντήλ, η οποία και αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κάποιες ε, τώρα τροπολογίες θα πρέπει να συζητηθούν σε σχέση με το πολιτικό πλαίσιο. Το κέριο θέμα εδώ είναι ποιο είναι το μήνυμα το οποίο εμεί θέλουμε να δώσουμε στην γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής μας. και σχετικά οι τροπολογίες που έχουν διατυπωθεί από τον κύριο Κατρούγκαλ και τον κύριο Σόλτ είναι κάπως παράξενες για μένα αλλά πιστεύω ότι ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της Επιτροπής μας έχει μάλλον μια διαφορετική άποψη για τα θέματα αυτά. Η τροπολογία για την δυνητική θεραπεία σοκ που είναι η τροπολογία 5 εγώ πρέπει να διαφωνήσω γιατί η δασμολογική προστασία είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλή και υπάρχει ήδη ανταγωνισμός. Επίσης και για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα θα είναι κάπως μακρόσο το μεταβατικό διάστημα. Αυτά λοιπόν είναι η αξιολόγησή μου των τροπολογιών και πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση το κύριο θέμα είναι ποιο οικονομικό μοντέλο θέλει να επιλέξει η Γεωργία και πιστεύω ότι εμείς πρέπει να προκρίνουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο που βασίζεται σε ανοιχτές οικονομίες και ανοιχτές εμπορικές σχέσεις και μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δίνω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, πρώτα απ' όλα τον κύριο, στον κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Υποστηρίζουμε την έκθεση αυτή, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην κατάσταση που επικρατεί τώρα στη Γεωργία. Και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί τις τελευταίες μέρες και δεν είναι σαφές αν θα παραμείνει η κυβέρνηση της Γεωργίας. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω πόσο προσεκτικά μας παρακολουθούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων είπαν ότι το ΕΛ, τη μεγαλύτερη ομάδα, δεν θα υποστηρίξει την εμπορική συμφωνία με την Γεωργία. Αυτό είναι ένα καθαρό ψέμα. Και υπάρχει και κάποιος λόγος γι' αυτό. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες ιδέες οι οποίες ε, διατυπώθηκαν από, τα, από τους συντηρητικούς και δόθηκε αυτή η λαθασμένη εντύπωση που άρχισαν να ρωτούν, αν το ΕΛΚ άλλαζε άποψη. Μας παρακολουθούν πάρα πολύ καλά. Η διαδικασία όμως αυτή χρησιμοποιείται για να σταλούν διάφορα λανθασμένα μηνύματα σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαταλείψει αυτήν την περιοχή. Έχουμε ένα πολύ καλό ιστορικό συνένεση για τη Γεωργία. Ελπίζω ότι θα το κάνουμε και στην περίπτωση αυτή τη Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Μόση, δεν είναι παρόν, ο Ντέβιτ Μάρτιν. Δυστυχώ, ο Σκιώδη μα δεν έχει μπορέσει να έρθει, αλλά μου είπε να εκφράσω την συμφωνία μα με την άποψη του Όλη Ρεν. Και θεωρούμε ότι είναι εδώ μια περαιτέρω ευκαιρία να πλησιάσει η Γεωργία με το ευρωπαϊκό εμπόριο και να εφαρμόσει το κράτος δικαίου και να έχει περικές περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες καθώς και για επιχειρήσεις της Ένωσης στην Γεωργία. Νομίζω ότι είναι λοιπόν κατάσταση σε γουιν και για τους δύο. Με βάση την εφταξία, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Γενικά λοιπόν συμφωνούμε με τις τροπολογίες και την άποψη του κυρίου Όλη Ρέν. Μάλιστα, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος και τον κύριο Λαντσβέρκης και οποιονδήποτε άλλο που θέλει να ακούσει ότι η ομάδα μας υποστηρίζει τη θέση αυτή, πρέπει να το ξέρει. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία που έχει η εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γεωργία δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία περί τούτου και ευχαριστώ τον εισηγητή για το ανοιχτό του πνεύμα και για όλη την εργασία του συμφωνούμε με το, τελική, με το τελικό του συμπέρασμα και με τις συμβιβαστικέ τροπολογίες και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουν γίνει δεκτές και οι δικές μας τροπολογίες. Παρόλα αυτά, όπως είπε πολύ σωστά και ο ίδιος, υπάρχουν μερικές τροπολογίες που δεν γίνονται ομόφωνα δεκτές και για μας και ούτε εμείς μπορούμε να τις δεχτούμε. Εκείνες δηλαδή που υπέβαλαν οι συνάδελφοί μας από την ΚΟΕ. Γενικά λοιπόν η στάση μας θα είναι γενικά θετική. Ευχαριστούμε πολύ από την ΚΟΕ ο κύριος Κατρούγκαλος. Thank you, Mr. Chair. Well, our reference uh, to the shock therapy uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, η στάση για την θεραπεία σοκ βασίζεται στο ότι όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σαν μοχλός για την εφαρμογή ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου που θα αμφισβητήσει το δικό μας κοινωνικό πρότυπο. Γιατί εμείς θέλουμε το εμπόριο να προωθεί με την ευημερία αλλά να εξαρτάται και από το κατά πόσον θα πρόκειται για ε, ανάπτυξη με βάση τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αν θα γίνεται σεβαστή και κοινωνική διάσταση. Και γι' αυτό εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις τροπολογίες που, κατατέ, κατέθεσα με τον κύριο Σόλτ για την χρονική πίεση και τους περιορισμούς που πρέπει να δεχτούμε για να εκφράσουμε την άποψή μας και γιατί δεν έγινε διαβούλευση με σημαντικούς ενδιαφερόμενους σε εκείνη τη χώρα. Επίσης ζητούμε η Γεωργία να σεβαστεί το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι απλώς να αγνοεί κάτι σημαντικό για μας την ευημερία του λαού και την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καζαντό από τους Πράσινους δεν είναι εδώ. Ο κύριος Δάρτμουθ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ε, επιστήσω την προσοχή στο σημείο α της ε, σύστασης Λέει ότι είναι μία από τις πιο φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία άλλη τρίτη χώρα. Μα αυτή είναι μια πάρα πολύ απλή εμπορική συμφωνία την οποία εμείς υποστηρίζουμε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα της πολιτικοποίησης του εμπορίου. έχει μια σαφή πολιτική ατζέντα αυτή η συμφωνία. Ξέρω ότι το ΕΛΚ με παρακολουθεί πολύ προσεκτικά. Είπατε ότι υπάρχει ενότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την Ουκρανία. Μα ζείτε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει ομοφωνία ούτε και για το θέμα της ε, Είναι η πολιτικοποίηση του εμπορίου που δεν πρέπει να συμβαίνει. Η άλλη ανησυχία μας είναι για την διεύρυνση. Μας ανησυχεί ότι αυτή η φιλόδοξη συμφωνία είναι μια πίσω πόρτα για την διεύρυνση. Το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα στις εκλογές του 2009 είχε στο μανιφέστο του ότι, δεν, ότι υποστηρίζανε την Γεωργία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξέρω από τον εισηγητή, ο οποίος είναι πρώην Επίτροπος για τη Διεύθυνση να μας πει τα εξής. Θα ήθελα, αν μπορεί να το πει, ότι αυτό δεν είναι αυτή η συμφωνία δεν είναι πρόδρομος της διαδικασίας προσχώρησης της Γεωργίας και δεύτερον δεν θα υπάρξουν καθόλου χαλαρώσεις στις υποχρεώσεις για προξενικές θεωρήσεις μεταξύ Γεωργίας και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να προερχόνται από την εμπορική συμφωνία και αν Υπάρχει ήδη τώρα κάποια χαλάρωση στο μέλλον. Δεν θα ζητήσουν αυτός και οι συναδελφοί του να υπάρξουν περαιτέρω. Αυτές είναι οι από τον εισηγητή. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό θέμα. Δεν είναι μια ουσιαστική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και ο εισηγητής του ΕΛΚ το έκανε σαφό, σαφές αυτό. Αυτή, σε αυτή την επιτροπή μπορείτε απλώς να κάνετε ότι ακούτε τους άλλους. Είναι ευγενικό. Μπορείτε να μην τα ακούτε, αλλά κάνετε ότι τα ακούτε. Η κυρία Λεπέα. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές που μόλις έγιναν δεν εξυπηρέτησαν καμία τίποτα. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο αποσυνδεδεμένη από τους λαούς που αποσυνδέεται και από τα αποτελέσματα των εκλογών. Μόλις γίνανε εκλογές, ε, τις είδαμε τα αποτελέσματα στις έδρες μας έτσι γενικώς και ορίστος, αλλά κανείς δεν κατάλαβε τι υπόθηκε. Ε, δεν είμαστε χαζοί και προφανώς και γνωστοποιούμε αυτή την κατάσταση στους λαούς μας και πρέπει προφανώς να οργανωθούμε σιγά σιγά και όσο γίνεται και πιο σύντομα να προετοιμάσουμε την προσχώρηση της Γεωργίας. Όμως η ευρωπαϊκή λαή είναι κατά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και ότι αν γινόταν οργανωμένο δημοψήφισμα σε κάθε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε νέα διεύρυνση η απάντηση θα ήταν όχι και μάλλον θα ήταν και μαζικά όχι. Δεν ακούσατε τον κόσμο που σας είπε ότι η διεύρυνση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία την έχουν μετανιώσει πικρά γιατί δεν είδαν κανένα πλεονέκτημα από την είσοδο αυτών των νέων χωρών πέρα από την μεγαλύτερο ανταγωνισμό και μάλιστα αθέμητο ανταγωνισμό γιατί προφανώς αυτές οι χώρες ε, κατά κάποιους ε, είναι το απόθεμα ε, εργατικών χεριών χαμηλού κόστους. Άρα θέμε του ανταγωνισμού για τους δικούς μας εργαζόμενους. Και συνεχίζεται λες και δεν τρέχει κάστανο. Υπάρχει και ένα παραμύθι βάτραχος που ήθελε να γίνει πιο χοντρός από το βόδι. Μα θα σκάσετε με αυτή την ε, κατάσχετη όρεξη που δείχνετε. Αυτή η ακόρεστη όρεξη δεν θα χορτάσει από τους λαούς που εμείς αντιπροσωπεύουμε εδώ και δεν έχουν οι λαοί την ίδια όρεξη με εσά. Εγώ σας συμβουλεύω λοιπόν να στραφείτε προς τους λαούς και να τους ακούσετε τι λένε, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε πια να συνεχίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση ενώ οι ευρωπαϊκοί λαοί θέλουν να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο. Θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάσμα, της οποίας η Ευρωπαϊκή, το, οποίο, το πρώτο θύμα θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς μεγάλη μου χαρά. Αυτός από την Κομισιόν. Εκ του ονόματος του ο οποίος δεν μπορεί να είναι παρόν, θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Μία διευκρίνηση πρώτα απ' όλα. Η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται ήδη προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όχι, ναι. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν αποτελέσματα θεραπείας σοκ, γιατί η Γεωργία είναι ήδη αρκετά φιλελεύθερη στην εμπορική της πολιτική ήδη και γι' αυτό πήραμε κάποιες συνειδητές αποφάσεις για μια φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου σε ό,τι αφορά την φιλελευθερωποίηση του εμπορίου και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε μετά από μια συζήτηση μαζί τους στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για το σεβασμό των κοινωνικών, του κοινωνικού κεκτημένου. Αντίθετα, η κυβέρνηση της Γεωργίας φτύνει πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική διάσταση των πολιτικών αυτών και αυτό φαίνεται και στο περιεχόμενο της συμφωνίας και θα μπορούσα να διαβεβαιώσω τους ε, βουλευτές που ανέφεραν για το θέμα των προξενικών θεωρήσεων ότι πουθενά στο κείμενο δεν αναφέρεται η φιλελευθερωποίηση και τις προξενικές Είναι μια διαφορετική διαδικασία που δεν συνάπτεται με τις εμπορικές πτυχές της συμφωνίας σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες πρόνοιες αυτής της συμφωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την δέσμευση της Κομισιόν θα σας κρατά πληροφορημένους σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Θα το πράξουμε αυτό και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για πληροφορίες και είμαστε απόλυτα στην διάθεσή σας. Αυτά. Ο εισηγητής και πάλι. Σας ευχαριστώ και θέλω ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ε, στεναρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις τους. Ξέρω ότι υπάρχει ευρεία, ίσως όχι ομόφωνη υποστήριξη για αυτή τη γνωμοδότηση που θέλουμε να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή κατεύθυνση της γεωργίας και την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου ανοιχτής οικονομίας και εμπορίου. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα σε σχέση με τη φύση αυτής της συμφωνίας, σε σχέση με την διεύρυνση από την κυρία Λεπέν και τον κύριο Μόζερ Κατά τη δική μου άποψη, η Κομισιόν έχει ήδη απαντήσει με ένα πιστικό και πλήρη τρόπο. Δύο μοναχα σημεία θέλω να δείξω εδώ. Δύο. Σε αυτού του είδους συμφωνίες δεν υπάρχει μια εξελικτική ρήτρα που να οδηγεί στην ένταξη εν καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα πρέπει να αναμίξουμε τα θέματα διεύνησης με εμπορικές συμφωνίες αυτού του είδους. Όλα αυτά πρέπει να συζητούνται χωριστά και η μία ενδεχόμενη της σύνταξη θα αντιμετωπιστεί χωριστά. Δεύτερον, για την χαλάρωση στο καθεστώς προξενικών θεωρήσεων και αυτό πάλι ένα χωριστό θέμα και αν χρειαστεί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά. Και ως πρώην Επίτροπος Διεύρυνσης και ως Ευρωπαίος πολίτης θέλω να πω ότι αν δείτε την κεντροανατολική Ευρώπη τις χώρες της Διεύρυνσης του 2004 και του 2007 μπορείτε να δείτε ότι ήταν μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας μια ειρηνικής, δημοκρατικής και οικονομικής μεταμόρφωσης. Αυτές οι χώρες λοιπόν δεν ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τα προβλήματα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης ήταν οι παλιές ευρωπαϊκές χώρες. Και εξάλλου τα Δυτικά Βαλκάνια όπου η πολιτική διεύνηση λειτουργεί ήδη και λειτουργεί ακριβώς ως σταθεροποιητικός παράγον και έχει οδηγήσει σε ειρήνευση και σταθεροποίηση σε αυτή την περιοχή που την είχε ρημάξει ο πόλεμος, αυτά δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις υποχρεώσεις του. Τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται σε, μια σταθερή τροχιά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική σταθεροποίησης κρατώντας τη Σερβία στο δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη μια κρίση στην Ουκρανία, δεν θέλουμε και άλλη κρίση στα Δυτικά Βαλκάνια ή τη Σερβία. Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν τις επιτεύξεις της πολιτικής διεύνησης παρά το γεγονός ότι είναι ένα θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί. Το επόμενο σημείο τώρα είναι η γνωμοδότηση για τα νέα τρόφιμα. Εδώ έχουμε 98 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Εγώ κοιτάζοντας είδα ότι 31 από αυτές τις τροπολογίες δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές. Το έχουμε συζητήσει αυτό μαζί και με την εισηγήτρια και ως εκ τούτου πήραμε την απόφαση να τις θεωρήσουμε μη παραδεκτές και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη συμβολή τους στη γνωμοδότηση και ιδιαίτερα τους σκιώδει εισηγητέ, διότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους σκιώδει επ' της γνωμοδότησης και ως αποτέλεσμα φτάσαμε σε μεγάλη συνένεση και ευρεία συμφωνία που ελπίζω πως όλοι θα μπορέσουν να στηρίξουν αύριο στην ψηφοφορία. Είχαμε ευρεία συμφωνία όπως αναφέρατε, εστιάσαμε στα θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είμαι πεπισμένη ότι τέτοια στοχοθετημένη προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική για την Επιτροπή μας, καθώς και η πιο χρήσιμη για την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή που πρέπει να ασχοληθεί με ένα σωρό θέματα. Το κεντρικό ζήτημα λοιπόν για την ΙΝΤΑ είναι η αντιμετώπιση των παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες. Η τοποθέτηση παραδοσιακών τροφίμων στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς γραφειοκρατία. Θα πρέπει να παραμείνει τελικά όσο γίνεται πιο ασφαλής για τους καταναλωτές εντός της Ένωση. Ακολουθούμε αυτή την αρχή σε όλες τις συμβιβαστικέ και μέσα από τη συνεργασία με τους σκιώδεις βελτιώσαμε νομίζω τη γνωμοδότησή μου από πολλές απόψεις. Ε, δεν θα πρέπει δε να ε, μάλλον θα πρέπει να τοποθετούμε στο επίκεντρο της γνωμοδότησης την αρχή της προφύλαξης αλλά και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής υψηλού επίπεδου. Ε, δεν θα πρέπει ούτε να γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας fast track. Δημοκρατικός έλεγχος της διαδικασίας θα γίνεται μέσω της ουσιαστικής δυνατότητας που δίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο να θέσει βέτο σε, στην εισαγωγή αυτών των νέων τροφίμων, καθώς και στην, να ανακαλέσει την εφαρμογή αυτών των νέων κανόνων. Δε, ε, αυξήσαμε δε τη διαφάνεια αυτών των νέων ε, κανόνων. Επιπλέον όλων αυτών των συμβιβαστικών, που είναι έξι τον αριθμό και που αυστηρά σχετίζονται με τις ε, δύο, τις διάφορες κοινέ αρμοδιότητες, θα αναφέρω τις ανησυχίες σε κάποιων, κρατών, κάποιων μελών που αφορούν θέματα όπως η τοκετοθεσία και ευχαριστώ τη Μαρίαν και τον Ζωζέ για αυτές τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Υπάρχει η θέση μου για την κατάλογο ψηφοφορίας και με στη διαθεσή σας αν χρειάζεστε πληροφορίες πριν από την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θέλουμε να λάβουν το λόγο εσείς, ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς και μόνο θέλω να πω ότι είχαμε μία συνάντηση με την κυρία Κίρτον Λάρλινγκ. Έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που μας ικανοποιούν πλήρως και έχετε δίκιο κι εσείς και η συγγήτρια υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που θα μπορούσαν να είναι λογικές αλλά θεωρούμε ότι δεν εμπίπτουν στα θέματα της Επιτροπής μας είναι θέματα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν είναι τροπολογίες οι οποίες συνάπτονται με το έργο της δικής μας Επιτροπής. Επομένως νομίζω ότι είναι σωστό να απορριφθούν αυτές τις τροπολογίες χωρίς να εκφέρουμε γνώμη για το περιεχόμενό τους που πολλές φορές μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ενδιαφέρουσες όπως παραγωγή για, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Αυτά είναι θέματα όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν σε άλλο πλαίσιο και όχι στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Μας φαίνεται λοιπόν πολύ καλό το ότι έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε κάποιες συμβασικές λύσεις που γενικά θα τις υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ η Έμα. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έχει κάνει για το θέμα αυτό. Δεν μπόρεσα να πάω στη συνάντηση των ε, συντονιστών, αλλά σας Ανέφερα ποια ήταν η θέση μου και νομίζω ότι την έχετε λάβει υπόψη. Θέλω να κάνω σαφές ότι θέλω να υπάρξει ένας ενισχυμένος ρόλος για την, τροφιμή, για την υπηρεσία τροφιμικής ασφάλειας. Έχω αντιρρήσει σε κάτι τέτοιο γιατί αυτό οδηγήσει σε περαιτέρω εμπόδια και γραφειοκρατία στη διαδικασία και θα υποσκάψει και το ρόλο αυτού του φορέα γιατί θα επανέλθουν και πάλι τα πολιτικά ζητήματα και κάποιοι πολιτικοί θα μπορούν να μπλοκάρουν κάτι το οποίο τεχνικά και επιστημονικά έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή, από την υπηρεσία αυτή. Εμείς θα πρέπει να ελέγχουμε σε πολιτικό επίπεδο αλλά τις τεχνικές και επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες. Επομένως, δυστυχώς, η ομάδα μου δεν θα υποστηρίξει την έκθεσή σας αύριο όχι επειδή είμαστε κακοί άνθρωποι και είμαστε κατά του ανοίγματο της αγοράς, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι δημιουργούμε περαιτέρω φραγμούς έτσι. Η Μαρίκε. Μαρίκε. Δεν μπορούσε η Μαρίκε να είναι παρούσα, οπότε εγώ θα αναφέρω ποιες είναι οι απόψεις της. Και φυσικά δεν είμαι εμπειρογνώμων για το θέμα αυτό. Η Μαριάν θα ήθελα να συγχαρεί την εισηγήτρια. Θεωρούν ότι οι συμβαστικέ λύσει έχουν βελτιώσει την πρόταση τη Κομισιόν. Υπάρχει μια σαφή διάκριση μεταξύ νέων τροφίμων που προέρχονται από χημικέ διαδικασίε και αυτών που έχουν να κάνουν παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρε που δεν είχαν ιστορία κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διευκολυνθεί η είσοδο στην αγορά των δεύτερων αυτών τροφίμων. Επίση, υπάρχει βελτίωση τη πληροφόρηση των καταναλωτών και τη διαφάνεια θα γίνονται δημόσιες οι αποφάσεις της Κομισιόν και οι κανόνες για τα νέα τρόφιμα με διάκριση για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες και άλλα είδη ούτως επίν νέων τροφίμων. Και θα πρέπει να υπάρχει σαφής ετικετοθεσία για την προέλευση και τη σύσταση των τροφών αυτών. Επίσης έχουν ληφθεί οι απαραίτητες μέρημνες για την ασφάλεια των τροφίμων αυτών που θα βασίζονται στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της Υπηρεσίας για την Τροφιμική Ασφάλεια ΕΦΣΑ. Και επίσης αναφέρεται ότι πρέπει να σεβόμαστε την αρχή της πρόληψης όταν πρόκειται για την πολιτική τροφίμων. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην καινοτομία και την πρόσβαση των καταναλωτών σε νέα προϊόντα, αλλά και συγχρόνω και την ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Πρέπει να παραμείνουμε επάγρυπνοι και να δούμε τα αποτελέσματα της αδειοδότησης και οι εκθέσεις αξιολόγηση. θα πρέπει να μας το καταδεικνύει αυτό και επίση για τι τροπολογίε οι οποίε δεν θεώρησαν ότι είναι παραδεκτές γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά μα αφορούν σημαντικά θέματα όπως είναι η κλωνοποίηση, νανοτεχνολογίες, τα προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία και η Μαρία Σαρνέ. θα τα υποστηρίξει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία που είχαμε. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα και του συμβιβασμού που έχει πετύχει. όμω γιατί μερικέ από τι τροπολογίε μα ε, απορρίφθηκαν λόγω μιας πολύ αυστηρής ερμηνείας του τι καλύπτεται και τι δεν καλύπτεται από το πεδίο που καθόρισε η σχετική επιτροπή. Για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από άλλους, για την 38 και την 66 θέλω να μιλήσω. Γνωρίζουμε ότι η πολλή γραφειοκρατία μπορεί να είναι απαράδεκτο βάρος, αλλά τα νέα τρόφιμα αξίζει τον κόπο να τα εξετάσουμε λεπτομερώς. Δεν έχουν όλοι τις πληροφορίες που χρειάζονται, την προέλευση, τη σύνθεσή τους, την διατροφική τους αξία, διατροφική τους αξία κτλ. Τροπολογία 38. Όσο για την 66, εκεί λέμε ότι τα νέα προϊόντα θα επιτρέπονται μόνο αν δεν βλάπτουν το περιβάλλον και τα ζώα. Ευχαριστώ. Μποβέ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε κατά την αρχή της συζήτησης ότι μερικές τροπολογίες απορρίφθηκαν, ιδίως οι δικές μας. Διότι δεν μπαίνανε, λέει, στο πεδίο, στη δικαιοδοσία της Επιτροπής μας. Ας μην το ξανασυζητήσουμε γιατί το συζητήσαμε με την Προεδρία πολλές φορές. Αλλά εγώ θεωρώ βασικό να πούμε ότι είμαστε Επιτροπή που μιλάει για το εμπόριο και θα μιλήσουμε για νέα προϊόντα που ήδη υπάρχουν σε μερικά τρόφιμα, νανομόρια που έρχονται από ξένες, από τρίτες χώρες. Παίρνω παραδείγματα για τα νανομόρια, μεταλλικά νανομόρια, τα Ιβάν, Ηνωμένε Πολιτείε, Νότια Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία. Αυτές οι χώρες δεν έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί μας, έχουν. Ενώ σήμερα η ΕΦΣΑ αναγνωρίζει δημόσια ότι δεν μπορεί, δεν ξέρει αν μπορεί να αναλύσει τα νανομόρια ούτε στη διατροφή ούτε στο περιβάλλον, τις επιπτώσεις τους. Και μόλις δημοσιεύτηκε μια έκθεση τον Ιούλιο του 2014 από το Κέντρο Ατομικών Δοκιμών και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών με χρηματοδότηση της Ένωσης που λέει για πρώτη φορά ότι δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις τους. Μου φάνηκε λοιπόν σωστό μια επιτροπή που ασχολείται με το διεθνές εμπόριο να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει λέγοντας ότι απαγορεύουμε την εισαγωγή νανομορίων στη διατροφή διότι δεν έχουμε κανέναν τρόπο να γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις τους. Και έτσι νομίζω ότι είμαστε στη δικαιοδοσία μας. Θα είναι σκανδαλώδες τους επόμενους μήνες η ιστορία αυτή θα γίνει σκάνδαλο με τα νανομόρια. Σήμερα το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να αναλάβει την ευθύνη του σε μια γνωμοδότηση που θα απαγόρευε αυτή την εισαγωγή. Δυστυχώς δεν κατορθώθηκε αυτό εφόσον οι τροπολογίες που το πρότειναν απορρίφθηκαν από την Κομισιόν ή από την Επιτροπή μας. Πράγματι λέει και ο πρόεδρος και εγώ είμαι σχετικά αυστηρός γιατί έχουμε αντιμετωπίσει συγκρούσεις με άλλες επιτροπές όταν μπαίνουν στα δικά μας χωράφια αυτές οι άλλες επιτροπές. Ακόμα λοιπόν και αν θεωρώ ότι είναι σωστές σε επίπεδο περιεχομένου αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να δούμε τι συνάπτεται με τα εμπορικά θέματα και όχι εσείς είσαστε μία αλεπού και έχετε τη δυνατότητα αυτές τις ε, τροπολογίες να τις και να τις ε, καταθέσετε σε άλλες επιτροπές ώστε να μην πάνε στράφη. Η κυρία Γκίνη. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του, την εισηγήτρια συγγνώμη. Ε, ε, ε, εδώ δεν έχουμε ιστορία σημαντική καταναλωτική. Είναι μια ανεπτυσσόμενη αγορά και μεγάλε ευκαιρίε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ωστόσο, πρέπει με προσοχή να ρυθμιστούν όλα αυτά για να αγγιηθούμε την ασφάλεια των καταναλωτών. Εμεί προσπαθήσαμε να δώσουμε περισσότερε κανόνε για τα τρόφιμα που έρχονται από τρίτε χώρε, που δεν υπόκειται δηλαδή στου κανόνε που έχουμε εμεί εδώ στην Ευρώπη. Και ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένα κατάλογο με όλα αυτά τα προϊόντα, αυτή να είναι δημόσια και να μπορεί κάθε πολίτης να τη συμβουλευτεί. Επιμείναμε επίσης σε περίπτωση προβλήματος για την ασφάλεια να μπορούμε εγκαίρως να απαγορεύσουμε την εισαγωγή αυτών των μη ασφαλών τροφίμων. Που προσπαθήσαμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα ε, πλαίσιο πιο ρυθμισμένο ε, για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των καταναλωτών. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που συμπεριέλαβε πολλέ από τι τροπολογίε μα τις κοινέ τροπολογίε. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία ανέφεραν ε, τα μέλη της Επιτροπής σας, ε, δηλαδή ε, τους ορισμούς, τον κατάλογο δηλαδή των ε, στοιχείων που θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κανονισμό. Στο αρχικό μας σχέδιο δεν υποβάλαμε κατάλογο προϊόντων ή ε, τροφίμων γιατί ε, πιστέψαμε πως έτσι θα μπορούσε να υπάρξει μια ευρύτερη εφαρμογή. Όμως κάποιοι κάποιες τροπολογίες δηλώνουν ότι θέλουν να επενεσεχθεί κατάλογος προϊόντων και ορισμός αυτών ε, μεταποιημένων ή μη μεταποιημένων είναι μια πρόταση που μπορούμε να δεχτούμε. Τώρα, τα κλωνοποιημένα ζώα. Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο μιας παράλληλης πρότασης γιατί η Κομισιόν θέλησε να ε, μιλήσει για αυτή τη συζήτηση για τα νέα τρόφιμα ε, γνωρίζοντας ότι η συζήτηση επ' αυτών και επί των προϊόντων αυτών θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη πολιτική σε φύση και σίγουρα πολύ μακρά. Ωστόσο, κατανοούμε πως υπάρχει ένα κενό που θα πρέπει να συμπληρωθεί ε, ανάμεσα στην παλιά ε, νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα που έλεγε ότι τα τρόφιμα που προέρχονταν από κλόνους ήταν νέα τρόφιμα και άρα έπρεπε να αξιολογηθούν από την ΕΦΣΑ και την μελλοντική νομοθεσία περί κλόνων που ε, προτείνει την απαγόρευση της κατανάλωσης του κρέατος του γάλακτος των κλωνοποιημένων ζώων. Καταλαβαίνουμε πως εδώ υπάρχει ε, ένα κενό για την ώρα και ε, άρα θέλουμε να καλυφθεί αυτό το κενό για τα τρόφιμα που προέρχονται από κλόνος να ε, θεωρηθούν νέα τρόφιμα. Κάτι και για τα νανοστοιχεία, μόρια. Έχουμε μια νομοθεσία για Έχουμε μια νομοθεσία που είναι πεπαλαιωμένη και προτείνουμε να αλλάξει. Προτείνουμε μια κατεξοδότηση πράξη στο προηγούμενο κοινοβούλιο και το προηγούμενο κοινοβούλιο είχε απορρίψει αυτήν την κατεξοδότηση πράξη διότι είχαμε προτείνει να αποκλειστούν τα πρόσθετα στοιχεία που υπάρχουν στην αγορά εδώ και δεκαετίες ε, αλλά προστάτευαν τα νανομόρια με μια κατεξιδότηση πράξη λαμβάνοντας υπόψη την θέση του προηγούμενου κοινοβουλίου που είχε απορρίψει την πρώτη ε, πράξη ε, και αυτό θα πρέπει να έρθει προς συζήτηση σύντομα στις επόμενες εβδομάδες. Γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε να έχουμε έναν ορισμό των νανομορίων σε ένα μονοκείμενο. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, ορισμούς σε δύο διαφορετικά κείμενα που θα, υπο, που θα υποστούν διαφορετικές εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και θα υποβληθούν σε διαφορετικούς ε, πυρογνώμονες για να έχουμε απόκληση των ορισμών. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει μια αντιστοιχισμένη αναφορά με τον ορισμό που υπάρχει στο κείμενο για την ετικετοθεσία. Επίσης υπάρχει το μεγάλο θέμα του κατοφλίου. Κατοφλίου δηλαδή και κατανομή για την διανομή. Θα πρέπει να... Συγγνώμη, κατανομή, αν πρέπει να πάρουμε 5%, 10% ή... Ωστόσο, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι πρέπει να πάρουμε το χαμηλότερο κατόφλι, δηλαδή το 10%. Το πρόβλημα είναι ότι οι τεχνικές διάγνωσης που έχουμε τώρα δεν επιτρέπουν να εντοπίσουμε 10% μορίων σε ένα συστατικό για την ώρα. Η επιστήμη είναι περιορισμένη σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό και προτείνουμε το εξή στοιχείο. Δηλαδή, να, το 50%. Αλλά μόλις θα εξελιχθεί η επιστήμη στο κατόφλι διάγνωση, ναι, είναι, είναι σοβαρή η πρότασή μου κύριε Μποβέ, ε, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ιδιαίτερα στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Όχι, δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε όλα, γιατί δεν ξέρετε πόσο έχει μέσα και δεν ξέρετε καν αν έχει μέσα, ούτε πόσο, ούτε αν. Δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε. Δηλαδή, εμπιστευόμαστε την επιστήμη γιατί είμαστε βέβαιοι ότι στο μέλλον θα εξελιχθεί το πράγμα και άρα θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε το κατόφλι. Έχουμε επίσης, μάλλον ε, στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ε, υπήρχε, υπήρχαν ε, συγκεκριμένες νομοθεσίες που υπήρχαν ήδη σε άλλες ε, νομοθεσίες και που δεν έπρεπε να βάλουμε σε αυτά τα κείμενα για τα νέα τρόφιμα συγκεκριμένες επιπλέον διατάξεις γιατί πρόκειται για επανάληψη νομική του τι ήδη υπάρχει. Είναι σαφές τόσο για την αρχή της προφύλαξης ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα εφαρμοστούν για τα νέα τρόφιμα. Η αρχή της προφύλαξης εγγράφεται ε, στην βίβλο για την νομοθεσία, το General Food Law, για περιτροφήμων και άρα δεν χρειάζεται να την εφαρμόσουμε. Για την συμφωνία αυτή εσείς προτείνετε η Κομισιόν να κάνει μια έκθεση πέντε χρόνια μετά από την θέση σε εφαρμογή αυτής της Έκθεση και παραμονή στο, γενικού, στο Γενικούλε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε δύο χρόνια στις επιχειρήσεις και τι τρίτες χώρες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και έτσι θα έχουμε μονάχα τρία χρόνια εφαρμογής που θα μπορούν να ληφθούν υπόψη σε μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι είναι μικρό το χρονικό αυτό διάστημα γιατί υπάρχει πάντα ο απαραίτητος χρόνος για την εφαρμογή. Θα προτιμούσαμε να έχουμε μια έκθεση όχι επί τη βάση πέντε ετών, αλλά και επί τη βάση περαιτέρω χρόνων. Η Κομισιόν υποστηρίζει καταρχήν το να κάνει εκθέσεις. Αλλά αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Και αυτά ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Βλέπετε ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι τελείως. Το τελευταίο θέμα για τις αναφορές, οι συμβιβαστικές τροπολογίες μιλούν για πέντε χρόνια μετά την θέση ενισχύ. Λάβαμε υπόψη λοιπόν τις ανησυχίες της Κομισιόν ως προς το θέμα των αναφορών. Ελπίζω μεγάλη πλειοψηφία να μπορέσει να στηρίξει την έκθεση και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Συνήθω δεν μπορεί να ικανοποιήσει κανείς όλο τον κόσμο, αλλά ευχαριστούμε για την προσπάθειά σας. Το θέμα είναι να ικανοποιήσετε στο δυνατόν περισσότερο. Πάμε στο σημείο 17 πλέον. Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζιγκαπούρης. Έχουμε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά αγαθά και υπηρεσίες που ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου 2013 έχει συμφωνηθεί και μετά εκ των υστέρων υπήρξε το τμήμα των επενδύσεων που έχει τύχει διαπραγματεύσεων και στις 16 Οκτωβρίου έκλεισε και αυτή η διαπραγμάτευση και επομένως έχετε στα χέρια σας τα αποτελέσματα της ε, διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε με αυτά τα πράγματα. Και επίσης ξέρετε ότι η Κομισιόν στις 30 Οκτωβρίου απεφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτήν την περίπτωση για να διευκρινίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πότε μια συμφωνία είναι μεικτή συμφωνία και πότε αφορά αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 207 της συνθήκης της Λισαβόνας. Mm. Και φυσικά αυτό είναι ένα πολιτικά λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Και χαίρομαι που ο κύριος διαπραγματευτής, ο κύριος Σλέγκμιχ, είναι μαζί μας και θα του δώσω το λόγο για να δώσω μετά το λόγο στον μόνιμο συγκεκριτή μας, τον κύριο Ντέιβιτ Μάρτιν. Αναπάντεχο, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος Είχαμε μια ομάδα επιτήρησης για αυτό το θέμα της Σιγκαπούρης και μετά τις διαπραγματεύσεις για πρώτη φορά από τότε που ε, εγκρίνεται η συμφωνία σήμερα δηλαδή έχω μερικά και απορίες η μία είναι ότι ξέχασα να πω νωρίτερα κάτι για την ασφαλιστική ρήτρα ως προς τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Ακούσαμε φήμες ότι η Κομισιόν ήθελε οριζόντια ασφαλιστική ρήτρα και για μελλοντικές συμφωνίες να καλύπτει. Δεύτερον, κάτι που το έθεσα στην ομάδα επιτήρηση, αλλά θέλω να το θέσω και εδώ, για το θέμα του εμπορίου ως βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι τελείως υπανάπτυκτη η κοινωνία των πολιτών στη Σιγκαπούρη και θα ήθελα να δω τι φρονεί από αυτού η Κομισιόν ώστε να είναι βέβαιο ότι η εντόπια συμβουλευτική ομάδα θα λειτουργήσει όπως πρέπει και έπειτα κάτι που δεν είναι καθαρά ευθύνη των διαπραγματευτών, αλλά υπήρξαν τελευταία εξελίξεις στη Σιγκαπούρη. Η μία είναι η επαναφορά της θανατικής ποινής και η άλλη κάτι πολύ φιλελεύθερα μέτρα για την ομοφιλοφιλία. Συνδέεται αυτό και πώς με την εμπορική μας συμφωνία. Μάλιστα πρέπει να τα βάλουμε στη σειρά. Υπήρχε η συμφωνία πλην την προστασία, της προστασίας των επενδύσεων και χρειάστηκε τόσος χρόνος για να τελειώσει η συμφωνία ακριβώς λόγω αυτού που είπατε ότι είναι πολιτικά ελεπτό το θέμα ευαίσθητο όχι μόνο για μας αλλά και για τους φίλους μας στην Σιγκαπούρη που προσπάθησαν να διασφαλίσουν ότι η διαπραγμάτευση θα είναι μοντέρνα και σωστή. Μοντέρνα. Και το αποτέλεσμα ήταν καλό, αν και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, τα θέματα που, που παρέμεναν λύθηκαν και αυτά και από πλευράς της Κομισιόν θεωρούμε ότι για τις επενδύσεις άξιζε τον κόπο η καθυστέρηση. Γιατί εδώ συμπεριλάβαμε σχεδόν, σχεδόν όλες, όχι όλες, όλες, αλλά σχεδόν όλες τις καινοτομίες καμιά δωδεκαριά, καμιά ντουζίνα χώρες μέλη έχουν και αυτές BITs που λέμε, Έχουμε αυτή τη στιγμή καλύτερο ορισμό τι είναι δίκαια μεταχείριση των επενδυτών και αποσαφηνίζουμε ότι δεν θα πρόκειται μόνο για τυπική αλλαγή αλλά για την ουσία του θέματος των περιουσιών. Επίσης υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες δεν μπορεί κανείς να επιλεκτικά να εφαρμόσει μία από τις συνθήκες εκείνες. Πλήρης σεβασμός των διαμεσολαβήσεων και των συμπεφωνημένων. Και έχουν ληφθεί όλα αυτά υπόψη λοιπόν, αν και δεν ήταν πάντα εύκολο να τους πείσουμε. ότι χρειάζονται καλύτεροι κανόνες για το μέλλον. Είναι εύκολο. Ας σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι αυτά είναι τα ουσιώδη. Να πω μόνο κάτι για τη διαδικασία είναι σαφές ότι οι προσπάθειες για μεγαλύτερη σαφήνεια και στις γνωμοδοτήσεις του συνεδρίου ή του δικαστηρίου ήταν από τους παράγοντες που καθυστέρησαν το αποτέλεσμα. Η καινούργια επιτροπή βέβαια πρέπει να αποφασίσει. Μέχρι τώρα έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα για θέματα μεταφορών, επενδύσεων και άλλων. Και ελπίζουμε στο μέλλον όλα αυτά να είναι πιο προβλέψιμα. Ολόκληρη τη συμφωνία την συζητούμε και δεν θεωρούμε ότι η αποσύνδεση των επενδύσεων από τα υπόλοιπα είναι κάτι το θετικό. Last year. I Ας σταματήσω, αλλά να απαντήσω και σε αυτά που είπε ο Δαβίδ Μάρτιν για την ρήτρα ασφαλεία, τη οριζόντια ημί, το έχουμε συζητήσει και πρέπει να ελέγξω, να επαληθεύσω αν ισχύει αυτά που ισχύουν, αν ισχύουν αυτά που ισχύουν για το ΑΣΕΑΝ ή αν γίνεται η ρήτρα ασφαλείας μεμονωμένα για κάθε συμφωνία όπως έγινε με την Κορέα και άλλες χώρες. Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει γίνεται ακόμα η εσωτερική συζήτηση. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχετε δίκιο διότι δεν θέλουμε ούτε οι άλλοι να μας πούνε ούτε εμείς να πούμε τι θα κάνουν με, τους, με τις δικές τους ε, συμβουλευτικές ομάδες. γιατί υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα σχολιασμού. Το όλο θέμα του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η συνεργασία και το θέμα του ποιος είναι ο συνομιλητής. Τέλος, για τις συμφωνίες εταιρικότητας, δεν είναι το σημερινό μας θέμα βέβαια, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να αποφανθούμε και επ' αυτού συνεργασία και εταιρική σχέση. Επίσης το θέμα που συζητούσαμε μέχρι τώρα για την διαφάνεια της φορολόγησης. Δεν υπάρχει διαφωνία, αλλά υπήρξαν διάφορες γνώμες σε μια καλή και σωστή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα είναι παρόν. Έμα. Και δάκρυα. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ στην απόφαση του δικαστηρίου που περιμένει η Κομισιόν. Είπε η Κομισιόν πρέπει να περιμένουμε για το πακέτο επενδύσεων για να προχωρήσουμε. Αλλά πόσο να περιμένουμε και μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το κείμενο το οποίο θα παρουσιαστεί έχει περάσει το νομικό έλεγχο και υπάρχει ως τελικό τελικό κείμενο και τι αντίκτυπο θα έχει στις άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου σε επίπεδο διαδικασίας. Λέτε ότι για τη Σιγκαπούρ θα πρέπει να περιμένουμε 12-15 μήνες. Τι θα γίνει με τις άλλες. Η Μαρέικε. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να μιλήσω για την διαδικασία επίλυσης διαμαχών μεταξύ κρατών και περιττών είναι η ίδια όπως στην περίπτωση συμφωνής με τον Καναδά ή όχι. Και σε σχέση με την προτινόμενη απόφαση που θα πρέπει να πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, περιμένετε να υπάρχει κάποια, κάποιος διαχωρισμός στη διαδικασία κύρωσης και πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Αν κάποια τμήματα πρέπει να κυρωθούν από τα κράτη-μέλη, από τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τα άλλα, μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θα σημαίνει κάτι τέτοιο και πώς αλλάζει αυτό τον σχεδιασμό σας. τι θα σημαίνει αυτό το να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και τα επόμενα ε, βήματα για την τελική ε, κύρωση. Κυρία Μίλλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανησυχούμε πάρα πολύ για αυτή τη διαδικασία ελευθερών εμπορίου, γιατί μπορεί να είναι η πρώτη φορά που εισάγεται η επίλυση διαμαχών μεταξύ κρατών μελών και επενδυτών. Αυτό είναι κάτι που έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες και υπήρξαν 150.000 συμβολές στη δημόσια συζήτηση. Ακόμα και ο κύριος Γιούνκερ δεν υποστηρίζει τα ιδιωτικά δικαστήρια <clears throat> ή τους διαιτητικούς μηχανισμούς που μπορούν να καταλήξουν σε καλά αποτελέσματα δεν χρειάζεται να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους. Η κυρία Μάστρομ είπε ότι θέλει να βγάλει το ISDS από τη συμφωνία TTIP. Γιατί να συνεχίζει αυτή την υποστήριξη σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης δεν μου αρέσει η ιδέα ότι ο κύριος Δεχούχ, το πρώην επίτροπος, έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ερμηνεύσει τη συνδίκη Λισαβόνα για το αν τα εθνικά κράτη μπορούν να παρα... παρεμβαίνουν σε αυτέ τι περιπτώσει. Ε, Συμφωνίε όπω η ΣΥΤΑ και η Τίτιπ, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν μια τέτοια αντιμετώπιση. Θα ακολουθήσει μια πορεία με τοπική σύγκρουση η κυρία Μάλστρομ ή θα αποσύρει την αίτησή τη ακούγοντα την άποψη του Κοινοβουλίου. <clears throat> Κύριος Δαρτμούθης. Όχι, περιμένω την κυρία να λάβει πρώτο το λόγο. Και εγώ επανέρχομαι στην ε, ρήτρα ε, ISDS και εδώ βλέπω ότι δίνεται η δυνατότητα στις πολυεθνικές να μιλήσουν για απώλειες, για ζημιές. Γιατί όμως αυτή η ρήτρα ε, που ισχύει για τις τρίτες χώρες ε, να μην ισχύει για τη Σιγκαπούρη που είναι ναι μικρή χώρα αλλά ε, είναι τόσο πλούσια που μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές άλλες ε, τρίτες χώρες. Μπορεί αυτό να στραφεί εναντίον μας εάν η Σιγκαπούρη δεν ε, επενδύσει πια στην... Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ασιατικός επενδυτής και πραγματικά με εντυπωσιάζει γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή, να, να ενταχθεί αυτή η ρίστρα SDS εδώ πέρα. Όμω να μην δώσουμε και υπερβολικά πολύ δύναμη στους ιδιώτες επενδυτέ, εδώ και σε άλλες ε, ε, συνθήκες. Οποιοδήποτε πολίτης δεν μπορεί να στραφεί σε ένα υπερεθνικό δικαστήριο για να στηρίξει τα δικά του δικαιώματα, γιατί τότε μια υπερεθνική, πολυεθνική να μπορεί να το κάνει. Um, Σα ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι το EISDS είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε την προστασία των, επενδύσεων ενώ εγγυόμεθα και το δικαίωμα νομοθέτησης. Ε, τώρα, αν η Σιγκαπούρη θέλει να θεσπίσει το τη μορφή των ε, ασιατικών συμφωνιών και δεν υπάρξει εξισορρόπηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ασιατικές χώρες, γιατί στο καλό πάντα μιλάμε μόνο για προστασία επενδυτών και δικαιώματα επενδυτών και δεν μιλάμε καθόλου για ευθύνε επενδυτών ταυτόχρονα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για, αν δούμε μάλλον τι άλλε χώρε που έρχονται στη σειρά από πίσω. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μιλάμε εδώ για μια σύνδεση με τον ΟΑΣΕ, ΩΣΑ ε, με τις ε, μη δεσμευτικέ ε, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά είναι το πιο μικρό μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση τουλάχιστον. Η Κομισιόν πιστεύει ότι μια από τις προσθήκες στην συμφωνία με την Σιγκαπούρη για τη δυνατότητα χρήσης ε, θεμητών προσδοκιών ως ε, το αιτιολόγηση ότι υπήρξε άδικη ή μη συμμεταχείριση ή απαλωτρίωση. Αυτό δημιουργεί παραθυράκι για αν όχι γιατί υπάρχει. Äh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω και πάλι Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε είναι το πρακτέον. Τι θα κάνουμε με αυτή τη διαδικασία διαμεσολάβησης και περιμένουμε το δικαστήριο να μας δώσει τα φώτα του. Ποια είναι η ασφάλεια που προκύπτει για μας όταν έχουμε μία εμπορική συμφωνία υπόπερνευστή της Σιγκαπούρης ότι δεν χρειάζεται το ISDS γιατί τότε δεν το αποχωρήσουμε από τη συμφωνία. Μπορεί να έχει διαφορετική άποψη κανείς για το αν πρέπει να υπάρχει ή όχι μια τέτοια συμφωνία. Αλλά εγώ δεν έχω πάρει καμία απάντηση γιατί η Κομισιόν μας λέει ότι είναι αδύνατο να αποσυνδέσει τα θέματα επενδύσεων από την εμπορική συμφωνία. Η Τζούλη επίσης αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορές με την αρχική συμφωνία. Ο χρόνος αυτός λοιπόν που θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες ΑΣΕΑΝ. Και τέλος, ποια είναι η θέση αυτής της συμφωνίας μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν ήδη κάποιες ε, εμπειρίες στα πλαίσια του ΠΟΕ που να δημιουργούν και ανησυχίες σε σχέση με μια τόσο πλήρη συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Εγώ θα ήθελα να γίνει σαφές ότι και σαφές τις χώρες με τις χώρες ΑΣΕΑΝ να λάβουμε υπόψη την πλήρη πολυπλοκότητα των προβλημάτων και τα κείμενα τα οποία έχω δει μέχρι στιγμής δεν με καλύπτουν για το θέμα αυτό. Ο κύριος Τσίκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, ε, για την ολοκλήρωση, για το συμπέρασμα μάλλον αυτού του κεφαλαίου που αφορά τις επενδύσεις, ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες νομικές φύσης παρατηρήσεις. Οι διατάξεις ε, αυτές περιλαμβάνονται σε διάφορες εμπορικές συμφωνίες, όμως μέχρι στιγμής οι χώρες δεν τις έχουν χρησιμοποιήσει. Γίνεται λόγος για απουσία διαφάνειας, για περιτές ε, ρήτρε κτλ. Εγώ θεώρησα σκόπιμο να κάνω μια ευάθυνση και να προβώ σε κάποιες ενδείξεις ε, υποδείξεις και επί τη βάση αυτών των παρατηρήσεων ε, διαπίστωσα ότι σχεδόν όλες οι περιπτώσεις ε, που λύθηκαν ε, με το ISDS έγιναν μέχρι το 591. Από το 51 και μετά μόνο 85 υποθέσεις επιλήθηκαν υπέρ των επενδυτών. Τα ποσοστά, μάλλον με ποσοστά σημαίνει ότι μόνο 15% των υποθέσεων τις έχασε το κράτος. Θα πρέπει αυτό όμως να το διευκρινίσουμε. Από τις 85 υποθέσεις προϋποθέσεις που κέρδισαν οι επενδυτές, το 75% είναι επενδυτές που επικράτησαν έναντι κρατών ε, της ε, Νότιας Αμερικής και του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ. Και αυτό το γεγονός δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί για γνωστούς και ευνόητους λόγους. Για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε μόνο 11 υποθέσεις όπου ο επενδυτής επικράτησε του κράτους. Ε, πρόκειται για Ευρωπαίους που ποτέ δεν έχασαν υποθέσεις κατά των κρατών ε, εκτός ε, ε, κράτη δηλαδή όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω πως θα μπορούσα έτσι να συμβάλλω, δεν θέλω να κάνω στήρακτη και ίσως θα έπρεπε να γίνει πιο τεχνική και νομική εμβάθυνση παρά ιδεολογική και πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κασπάρη ο τελευταίος ομιλητής. Και εγώ θέλω να μπω στο θέμα των ε, και Ε, επενδύσεων, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν μιλήσει για τον, την αποσύνδεσή του. Αλλά είχαμε μία εντολή διαπραγμάτευσης, υπενθυμίζω, που είχε σε στόχο να αντιμετωπίσει όλες τις χώρες ΑΣΕΑΝ και υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες χρειάζονται για εσωτερικούς λόγους μια συμφωνία για τα επενδυτικά θέματα και θα ήθελα η Κομισιόν να μας εξηγήσει στις επόμενες εβδομάδες πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε το θέμα της προστασίας των επενδυτών στη σύμφωνία με την Σιγκαπούρη. και πώς η Κομισιόν μας έχει δώσει τις εκθέσεις που έχει ζητήσει πάντα το Κοινοβούλιο για τη συμφωνία αυτή, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια άποψη για το, την τελική απόφαση και συγχαίρω την Κομισιόν που θα πάει ενώπιον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριου για την υπόθεση αυτή. Θα πρέπει όμως να βιαστείτε. Το θέμα αυτό θα πρέπει να διαλευκανθεί το ταχύτερο δυνατό. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που είναι απαραίτητα ώστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να έχει σχετικά γρήγορα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να μπορέσει να καταλήξει σε μια απόφαση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό και για μελλοντικέ συμφωνίες ελευθερών εμπορίου δεν είναι η εντύπωσή μου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αφαιρέσει εξουσίες από τα Εθνικά Κοινοβούλια, μάλλον το αντίθετο πιστεύω ότι θέλει να δώσει αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω στα εθνικά κράτη με το άρθρο 207. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω διευκρινήσει. και είναι απαραίτητο φυσικά όπως ελέγχθη να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε το κείμενο της Κομισιόν για την εμπορική αυτή συμφωνία σε σχέση με το θέμα αυτό που θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πότε θα έχουμε το κείμενο αυτό λοιπόν? Ευχαριστώ πολύ λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να προσπαθήσω να απαντήσω όσο με, μου επιτρέπει ο Γιαραμπής στα ερωτήματα αυτά και είναι και θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και η νέα Κομισιόν. Τι σημαίνει τώρα η διαδικασία αυτή κύρωσης για τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Αλλά ο Καναδάς ακόμα δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Πρέπει να κάνουμε την νομικό έλεγχο και τις μεταφράσεις και αν είναι 18 μήνες το χρονικό διάστημα που χρειάζεται τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά αλλά η Νέα Κομισιό θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά πώς να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Το κείμενο υπάρχει, είναι στην ιστοσελίδα μας και έχει αποσταλεί και στην Επιτροπή σας τη μέρα που τελειώσαμε τις διαπραγματεύσεις. Ο νομικός έλεγχος γίνεται κανονικά αλλά δεν περιλαμβάνει αυτό το κεφάλαιο. Συνεχίζεται μαζί με τους ε, Σίνκα Πουρέζους ο έλεγχος. Mm. Για το ερώτημα της κυρίας Σάκε για τη διαφορά μεταξύ της ΣΥΤΑ και της ε, συμφωνίας με τη Σιγκαπούρα. Σιγκαπούρη. Αυτό έχει να κάνει με την, ε, τις οδηγίες για τα χρηματοπιστωτικά. Εδώ υπήρχε μια σαφής συνένεση ότι στην περίπτωση του Καναδά οι ρυθμιστές ήταν σε θέση να λάβουν υπόψη όλα τα προβλήματα και αυτό βέβαια δεν ισχύει κατά ανάγκη με τη Σιγκαπούρη και εν πάση περιπτώσει όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα είχε κλείσει αυτό το ζήτημα και κανείς δεν ήταν έτοιμος να ξανανοίξει αυτά τα θέματα διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι όμως η κύρια διαφορά που θέλω να τονίσω αν συγκρίνεται τα κείμενα αυτά. Οι άλλες καινοτομίε που έχουμε ακούσαμε και από τον κύριο Κασπάρη ότι υπάρχει μία ε, εντολή για συνολικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Πιστεύω ότι είναι μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ε, διαβουλεύσεις που έχουμε για τη συμφωνία TTIP. Ζητήσαμε να μας δώσουν απαντήσεις για συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το τι πρέπει να πράξουμε εναπόκειται να δούμε κάποια, ποια από αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τη γενική μας πολιτική και ποια είναι θέματα που είναι ειδικά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω συγκεκριμένων ε, κινδύνων ή της διαφορετικής νομικής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτείων που μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτή των άλλων εταίρων μας. Αναφέρθηκε και το ερώτημα ότι η Σιγκαπούρη δεν είναι ένα της κυρίας Μίλλερ, η Σιγκαπούρη δεν είναι <clears throat> ένα ασταθές νομικό πλαίσιο. Το να υπάρχουν κανόνες για τους επενδυτές δεν είναι θέμα μονάχα σταθερού νομικού mm. πλαισίου, αλλά και διεθνών κανόνων και αν θέλουμε να τους εφαρμόσουμε και σε ποιο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, αν θεωρείτε ότι για, τη Σιγκαπούρη δεν θα χρειαστούμε τίποτα, τα μεγάλα κράτη-μέλη δεν ξέρω ποιος έθεσε αυτό το ερώτημα, αλλά κάποιος έκανε αυτό το σχόλιο. Πρέπει να επανέλθουμε στους αρχικούς κανόνες. Αν κάποιος θέλει να εναγάγει τα κράτη βάσει των τωρινών κανόνων μπορεί να το κάνει. Οποιοδήποτε επενδυτή μπορεί να το κάνει αυτό. Οι κύριες χώρες λοιπόν, οι οποίες επενδύουν ή παίρνουν επενδύσει από τη Σιγκαπούρη, καλύπτονται ήδη από προηγούμενε ε, συμφωνίες για επίλυση διαφορών. Τώρα για τις υποχρεώσεις των επενδυτών. Σίγουρα δέχομαι ότι δεν έχουμε μια απόλυτη ισοτιμία γιατί οι υποχρεώσεις των επενδύσεων είναι όλο το νομικό πλαίσιο που πρέπει να αποδεχτούν όταν πηγαίνουν σε μια χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κοιτάμε τα θέματα αυτά γιατί ακούμε τις εκκλήσεις που γίνονται και τις ε, κατευθυντήρες γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε. Θα εξετάσουμε και στο μέλλον γιατί καταλαβαίνουμε μπορεί να έχει νόημα να θέσουμε λίγη περισσότερη έμφαση στα θέματα αυτά ακόμα και αν είναι δυνατόν να ενισχύσουμε περισσότερες κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες όπως ξέρετε δυστυχώς δεν έχουν διεθνή οικουμενική κάλυψη και δεν είναι σε όλες τις χώρες. Κάποιες χώρες τις ακολουθούν, άλλες πάλι όχι. Ναι, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα για τα δικαιώματα που έχουν οι επενδυτέ και μπορούμε να εξετάσουμε και περαιτέρω ιδέες. Και ετέθηκε το θέμα των προσδοκιών. Νομίζω ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς κάνουν σαφές ότι η βασική ιδέα που τη διατρέχει είναι το pacta sunt servanda, ότι πρέπει να τηρούνται συμφωνίε και τα κάτι μελη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κυριαρχική του ε, δύναμη για να τι ανατρέψουν. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με μια προσδοκία να υπάρχουν συγκεκριμένα κέρδη, αλλά απλώ ότι μια κυβέρνηση πρέπει να μπορεί να δει τη διαβεβαιώσει ότι οι δεσμεύσει που έχει κάνει εναντί μια επενδυτική προσπάθειες θα τηρηθούν. Τα βλέπετε αυτά λοιπόν και στο νέο κείμενο όπου αναφερόμαστε για την διαφορά των απόψεων αυτών σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο νομικό κόσμο και στο εθνικό διεθνές δίκαιο που μπορούν όλα αυτά να δημιουργήσουν προβλήματα. Δύο λόγια για τα υπόλοιπα θέματα τώρα. Ναι, προφανώς κύριε Σούλτζε, πραγματευόμαστε το μεταξύ. Ε, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία ε, είναι σε αναμονή, αλλά πρέπει να δούμε και το περιφερειακό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε ανάμεσα στις όλες τις χώρες, γιατί και να τους πούμε ναι, ε, αρκετά καλό είναι το νομικό σας σύστημα, αλλά να πούμε μετά στην διπλανή χώρα ότι α, εσείς δεν είστε και πολύ καλοί, είστε δευτεροκλασσάτοι πολίτες και με εσάς δεν διαπραγματευόμαστε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στην προσέγγισή μας και να πούμε ότι εδώ έχουμε ε, τρία ότι, ότι πρέπει να δούμε μάλλον τι ε, γίνεται σε ολόκληρη την περιοχή κάθε φορά. Για να σας χαροποιήσω λίγο από την αμερικανική πλευρά έχουμε στατιστικές που λένε ότι με, σύμφωνα με την ΑΦΤΑ και τα αμερικανικά ε, καθεστώτα ε, υπάρχουν 55 ε, ISDS και 17.000 υποθέσεις στην ίδια περίοδο. Αυτό σας λέει ότι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις διώκονται δεν είναι και τίποτα το νέο. Συμβαίνει διαρκώς. Αλλά αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι μέσω αυτών των διεθνών υποχρεώσεων να δημιουργήσουμε περισσότερα δικαιώματα για τον εξωτερικό επενδυτή από ό,τι δίνουμε στους ίδιους τους πολίτες μας. Αν δείτε το κείμενο της Συμφωνίας ΣΥΤΑ έχουμε τουλάχιστον μια αρκετά καλή μελέτη από τη Γερμανία που λέει ότι η ΣΥΤΑ λέει λιγότερα ε, δικαιώματα στους ξένους επενδυτές από ότι στους πολίτες μας. Οπότε οι ξένοι επενδυτές ε, θα χρησιμοποιούν πάντοτε τα ε, χώρια δικαστήρια πριν στραφούν στα διεθνή. Έχουμε πάρει διάφορα κείμενα από την ε, έκθεση ε, για τη Σιγκαπούρη και για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα όσα ακούμε εδώ. Μία τελευταία ερώτηση αφορούσε γενικότερα το κείμενο νομίζω. Ναι, μάλιστα το κείμενο της δικαστικής υπόθεσης ε, νομίζω θα πάρει 4 με 8 εβδομάδες από ό,τι μου είπανε. Αλλά δεν θέλω βέβαια να το σας τορκιστώ, γιατί μου το είπαν απλώς. Ε, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Πάντως έχουν κάπως επιταχυνθεί τα πράγματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα. Ευχαριστώ, Ντέβιν. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Κυρίες και κύριοι, Έχουμε ένα πρόβλημα τώρα και το να καταγραφεί στα πρακτικά ή θα συζητήσουμε στα αγγλικά τις ομάδες παρακολούθησης, θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση αυτή. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε. Τι θέλετε, να το αναβάλουμε. Να προχωρήσουμε. Στα αγγλικά μονάχα.